We Να ξεκινήσουμε παρακαλώ. Να ξεκινήσουμε την πρωινή συνεδρίαση. Μια πρωινή και μια απογευματινή συνεδρίαση πολύ φορτωμένες με θέμα πολύ ενδιαφέρον την εξωτερική πολιτική ασφάλειας με εισηγητή τον κύριο Τζαμπάσκι, τον οποίο ευχαριστώ ιδιαίτερος, διότι υπέβαλε σχέδιο έκθεση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που είναι καθήλυνα αρμόδια και νομίζω ότι θα είναι πρωτοποριακό η Επιτροπή μας να έχει συζήτηση για το θέμα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, διότι πλέον νομίζω όλοι έχουμε κατανοήσει αυτή την έννοια, αλλά πρέπει να ενισχύσουμε κατά την πολιτική, πολιτιστική διάσταση στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και για να προλαμβάνουμε τις συγκρούσεις αλλά και για να προωθήσουμε την δυνατότητα να υπάρχει διαπολιτιστικός διάλογος και να ενισχυθούν οι διαπολιτιστικές διεθνείς σχέσεις. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Τζαμπάσκι, να θυμίσω ότι μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίε ω τι 21 Μαρτίου στι 5 το απόγευμα και ότι η ψηφοφορία στην Επιτροπή μα θα γίνει στι 26 Απριλίου, ενώ η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΑΦΚΟ στι 24 Μαου. Κύριε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την Γραμματεία της Επιτροπής Πολιτιστικών Υποθέσεων για την ε, βοήθειά τους στη σύνταξη της ε, γνωμοδότησης αυτής και για τις διοικητικές διευθετήσεις που επέτρεψαν να γίνουν. Με συγχωρείτε με τα γερμανικά υπάρχει πρόβλημα. Α, με τα αγγλικά. Τώρα. Ο ήχος. Δοκιμάστε παρακαλώ. Ο χρόνος που είχα στη διάθεσή μου για να συντάξω την έκθεση ήταν πολύ περιορισμένος. Ο η συγητή τη καθήλυνα αρμόδια επιτροπή, ο κ. Μπροκ, αρνήθηκε να επαναπρογραμματίσει την ψηφοφορία για να έχουμε περισσότερο χρόνο να εκφράσουμε τι απόψει μα. Ωστόσο, ο αρμόδιο τη επιτροπή μα από την γραμματεία κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία με του μεταφραστέ και μα δόθηκαν πέντε επιπλέον ημέρε για να μπορέσουμε να εκφράσουμε σωστά τις απόψεις, απόψεις μας. Η μετάφραση σε όλες τις γλώσσες ήταν έτοιμη την περασμένη Πέμπτη και ελπίζω ότι και άλλοι σκιώδεις εισηγητές θα μπορέσουν να μελετήσουν επαρκώς την έκθεση. Επιτρέψτε μου να παρουσιάσω εν συντομία τα εξή. Η ετήσια έκθεση της κυρίας Μογκερίνη για την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλεια το 2014 δεν αναφέρει τον όρο πολιτισμός. Θεωρούμε ότι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να προλαμβάνονται ε, οι ένοπλες συγκρούσεις και να προάγεται η ειρήνη. Αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα. Το άλλο ερώτημα είναι πώς αυτό θα μπορούσε να γίνει πράξη δεδομένη της αρμοδιότητας των κρατών μελών και τις αποφάσεις που μπορούν να λάβουν στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τη Συμφωνία των 28 κρατών ή ε, πολιτικοί ηθήνοντες μόνον. Μόνο έτσι μπορεί να ληφθεί η απόφαση εφόσον υπάρχει συνένεση. Εδώ λοιπόν μπορεί να υπάρχει σοβαρό ρόλο για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό στην ε, πολιτιστική διπλωματία. Αυτή θα είναι η δύναμη τη Ένωση και θα πρέπει να τονωθεί προκειμένου να προστατεύσουμε την πολιτιστική μα κληρονομιά. Επίση αυτό είναι ένα εργαλείο για να ενισχυθεί η ειρήνη, ο διαπολιτιστικό διάλογο και η σταθερότητα. Η έκθεση αναφέρεται και στο ρόλο του αθλητισμού Επίσης, αναφέρει την ιδέα ότι οι τρίτες χώρες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε βασικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του πολιτισμού και της παιδείας. Θα υποβάλω τροπολογίες για να αναπτύξω περισσότερο τη διάσταση του αθλητισμού και θα φροντίσω να γίνουν και πολλές, κάποιες προσθήκες ορισμένους παραγράφους. Ξέρετε ότι υπάρχει περιορισμός στους χαρακτήρες που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει και δεν μπορούν να ανακαλυφθούν όλα. Θα ήθελα λοιπόν να σας στείλω τις τροπολογίες μου σήμερα το απόγευμα ώστε να μπορέσετε να τοποθετηθείτε. Και θα προσπαθήσουμε να βρούμε, να καταλήξουμε και σε συμφωνία με του κοιόδη εισηγητέ. Όπω είπε και η κυρία Κώστα, η προθεσμή για την υποβολή των τροπολογιών είναι η Δευτέρα 21 Μαρτίου. Σημαντικό αυτό γιατί είναι και τα γενέθλιά μου. Με μεγάλη λοιπόν χαρά θα περιμένω να δω τις απόψεις των συναδέλφων. Μάλιστα, παρά το λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, θα παραμείνει ουσιώδης η έκθεση που συντάσσεται με την συμπερίληψη των απόψεών μας. Να θυμίσω για την πρώτη σας παρατηρήση αυτό που είπατε για την έκθεση για το 2014 Όντω, ο όρο του πολιτισμού δεν αναφέρεται. Είναι μια έλλειψη, αλλά εντοπίστηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζουμε ότι θα διορθωθεί αυτό με μια νέα εξισορρόπηση που θα συμπεριλαμβάνει και την πολιτική διάσταση. Και τώρα λόγο στους κοιόδης εισηγητέ, εφόσον βρίσκονται εδώ. Παρακαλώ κυρία Τρούπαλ. Ναι, ευχαριστώ για την παρουσίαση. Θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποια πράγματα που ήδη αναφέρατε και αυτό ότι στην διακρατική συνεργασία βάσει του πολιτιστικού διαλόγου ε, ο ρόλος του διαλόγου αυτό είναι πολύ σημαντικός για να προλαμβάνουμε την, ε, τις εχθροπραξίες και να ε, σταθεροποιείται η ειρήνη. Αυτή είναι μια στρατηγική προσέγγιση στην όλη διαχείριση των εξωτερικών μας σχέσεων διότι πρέπει να έχουμε μια καλύτερη, μεγαλύτερη έμφαση στην πολιτιστική διάσταση και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει. Όσο για την έκθεση του 2014, όντω ο πολιτισμό δεν αναφέρεται, αλλά ξέρετε, είχαμε αυτή την πρωτοβουλία του More Europe, τη περισσότερη Ευρώπη, και κατέστη σαφέ ότι θέλουν και ο πολιτισμό και η πολιτιστική διπλωματία να φανούν ε, σε ένα ισότιμο επίπεδο, να προβληθούν και να προχωρήσουμε με διάφορε οργανώσει και οργανισμού σε πολιτιστικά προγράμματα. Δηλαδή περισσότερο στο επίπεδο των μη κυβερνητικών οργανώσεων και τη κοινωνία των πολιτών είναι σημαντική η διάσταση αυτή, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να έχουν πλέον δυνατότητε να εκφραστούν, να έχουν συναλλαγέ μεταξύ του και διάλογο. Είναι λοιπόν στρατηγική σημασία να βεβαιωθούμε ότι ο πολιτισμό θα είναι ένα απόσπαστο τμήμα των ε, εξωτερικών πολιτικών και των πολιτικών ασφάλεια. Όπω για παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία, το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και εδώ, χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες πραγματικές δεσμεύσεις σε διμερή, και διακρατικά προγράμματα συνεργασίας με πολιτιστικά στοιχεία ή πολιτιστική διάσταση. Το συζητάμε συχνά αυτό, αλλά αν δούμε τη συμφωνία συνεργασίας, διαπιστώνουμε ότι ο ρόλος του πολιτισμού και της παιδείας δεν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο όσο θα θέλαμε εμείς. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια αλλαγή. Ευχαριστούμε. Συμφωνώ πολύ η κυρία Μπίλτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, τον κύριο Τζαμπάσκη, για την σύνταξη της έκθεσης αυτής που είναι πραγματικά στατική σημασία. Πράγματι είμαι πεπισμένη ότι η πολιτιστική διπλωματία μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο στην τήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας. Συμμερίζομαι τις απόψεις σας όταν μιλάτε για την ανάγκη να βασιστούμε σε διακυβερνητικές ε, μορφές συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα, αλλά θα πήγαινε ακόμη πιο πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κερδίσει αν έχει διάφορες στρατηγικές εταιρικές σχέσεις που ε, κατά τη διάρκεια τη ιστορία είδαμε να ωφελούν τα κράτη-μέλη και τις τρίτε χώρε. Σκέφτομαι ιδιαίτερα τι προνομιακέ σχέσει με τι χώρε τη Αφρική και να πω ότι η ίδια συμμετέχω στην αντιπροσωπεία των χωρών ΑΚΕ και ε, υπήρχε, προβλέπεται επίσκεψη στη Μαδαγασκάρη σύντομα με την οποία έχω καθέσει εδώ και χρόνια. Να ενισχύσουμε λοιπόν την εξωτερική πολιτική, ε, στην εξωτερική πολιτική διάσταση αυτή, ε, στη σχέση μας με διάφορα κράτη. Υπάρχει πολιτιστικός πλούτος που μπορεί να ωφελήσει την πολιτική μας και γι' αυτό θα ήθελα να επικεντρωθούμε στην παράγραφο 4 του, της έκθεσης που μιλάει για την προστασία των ε, ιστορικών πολιτιστικών μνημείων. Η διπλωματική μας ε, δραστηριότητα θα πρέπει να είναι φιλόδοξη. Είναι σημαντικό να εντοπίσουμε την καταστροφή των πολιτιστικών μνημείων στην Ευρώπη και στον κόσμο και να κοιτάξουμε πώς θα την προλάβουμε. Ε, η καταστροφή τη πολιτιστική κληρονομιά ε, σκοπεύει να καταστρέψει του ίδιου λαού, τη μνήμη του και την ιστορία του. Τα κάτι μέλη θα πρέπει να εντείνουν τη συνεργασία του στον τομέα αυτό, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι η πολιτιστική κληρονομιά των λαών, ιδίω τη Ευρώπη, δεν θα καταλήξουν το σκοπίδο την τη ιστορία ε, προ όφελο του πολιτισμού και τη παιδεία που θέλουμε να προστατεύσουμε. Έτσι λοιπόν αυτή η πολιτική διάσταση πρέπει να διέπει τις εξωτερικές μας σχέσεις και αυτό θα πρέπει να εντοπιστεί ε, και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να αξιοποιηθεί η προβολή και η απήχηση των ευρωπαϊκών πολιτιστικών κληρονομιών. Όσο για την παράγραφο 8 έχω κάποιες ε, επιφυλάξεις. Η Ελλάδα εδώ και ένα χρόνο λόγω χάρη δεν λαμβάνει κονδύλια από το πρόγραμμα Erasmus ε, Plus. Μου φαίνεται λοιπόν δύσκολο να αρχίσουμε να επεκτείνουμε το πρόγραμμα αυτό ε, σε τρίτα κράτη ήδη από τώρα, ενώ δεν έχουμε καλύψει τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Επίσης, πολλές καλές ιδέες δίνονται και σε άλλες παραγράφους της έκθεσης και ε, οι τροπολογίες μου ελπίζω να εμπλουτίσουν τις ε, εύστοχες αυτές προτάσεις και να έχουμε μια πραγματιστική και φιλόδοξη διατύπωση της πολιτιστικής μας διπλωματίας. Ευχαριστούμε, συνάδελφος Νέκοφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Τζαμπάσκι για τη δουλειά του στην έκθεση αυτή. Στηρίζω την ε, έκθεση του και συμφωνώ ότι δεν είναι θετικό στοιχείο ο πολιτισμός και η πολιτιστική διπλωματία να μην αναφέρονται στην ετήσια έκθεση για την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλεια. Είδαμε άλλωστε μόλις τα τελευταία χρονιά πόσο σημαντική είναι η διάσταση του πολιτισμού και της παιδείας. Κάτι άλλο σημαντικό είναι να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για τη συνεργασία και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς παγκοσμίω. Πρέπει να ληφθούν μέτρα κατά της εμπορίας πολιτιστικών αγαθών που μπορεί να αποδυναμώνουν την πολιτιστική κληρονομιά. Πρέπει να δημιουργηθούν ευνοϊκοί όροι για την ανταλλαγή δεδομένων και τη συνεργασία σε εμπόλεμες περιοχές, λόγου χάρη με τη λεγόμενη γαλάζια ασπίδα και τη στρατηγική της. Επίσης, πρέπει να συλλέξουμε στατιστικά δεδομένα στον ε, τομέα του πολιτισμού και για τον πολιτιστικό κλάδο γενικότερα που θα μας δείξει πώς ε, μπορούμε να προάγουμε την κοινωνική ευημερία τους καλλιτέχνες, όσους εργάζονται στην ε, βιομηχανία του πολιτισμού εντός εισαγωγικών, τον πολιτιστικό κλάδο. Δηλαδή, να ενθαρρύνουμε το διαπολιτιστικό διάλογο με διάφορες πρωτοβουλίες. Υπάρχουν ένα-δυο στοιχεία στα οποία θα επικεντρωθώ ως σκιώδης εισηγητής. Ε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υπογραμμίσω πόσο επιτυχημένες ήταν οι αντιδράσει μα για την πολιτιστική διάσταση στα πλαίσια τη κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό ο πολιτισμό για την ανθρώπινη εξέλιξη και γι' αυτό καλωσορίζω την πρόταση τη Επιτροπή που περιμένουμε τον Απρίλιο φέτος επί του θέματος. Ο πολιτισμός είναι πολύ σημαντικός για την εξωτερική πολιτική, διότι είναι ένας τρόπος να ενθαρρύνουμε το διαπολιτιστικό διάλογο. Και αυτός είναι ο λόγος που ο πολιτισμός θα πρέπει να είναι μέρος των αναπτυξιακών μας προγραμμάτων. Γι' αυτό θα πρέπει ε, η παιδεία και ο πολιτισμός να λάβουν μια πιο προεξαίχουσα θέση στην διατύπωση των στόχων μας. Πρέπει να συνεργαστούμε και με την UNESCO. Προκειμένου να βελτιωθεί η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και UNESCO πρέπει να εργαστούμε έξω από την προπατημένη. Δεν μπορούμε να παραμένουμε στη συνεργασία σε μερικά μόνο προγράμματα. Πρέπει να βαθυνθεί η συνεργασία μα σε θέματα παιδεία και πολιτισμού μακροπρόθεσμα. Γι' αυτό χρειάζεται ένα ετήσιο τυραφωμένο διάλογο υψηλότατου επίπεδου, προκειμένου να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αυτού του είδου τι προκλήσει. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι το θέμα είναι άκρο σημαντικό και δίνει και πολλές προοπτικές για το μέλλον. Υπόθηκαν ήδη πολλά, ιδίω από την Αντιπρόεδρο Τρούπελ και συμμερίζομαι απολύτω τι απόψει τη ότι πρέπει να δώσουμε μια στρατηγική διάσταση στο όλο θέμα με σημαντικά βήματα όπω τα τριετέ ε, πιλωτικό πρόγραμμα More Europe ή ε, αυτά που αναφέρει η προηγούμενη εκθέση μου για το θέμα αυτό. Για την ε, πολιτιστική πολιτική στην εξωτερική μα διπλωματία. Βλέπω ότι η συνάδελφο Γκριμπάτσκα θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να μιλήσω για την παράγραφο 8 και να την υπερασπιστώ. Θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Erasmus Plus, Erasmus διότι δεν μπορούμε, δεν θέλουμε να αποδυναμωθεί το μέσο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα από την σκοπιά των σχέσεών μας με τις τρίτες χώρες. Ευχαριστούμε για την συμβουλή και τη σύσταση αυτή. Ε, πριν σας ξαναδώσω το λόγο, θέλει μήπως το λόγο Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει κάποιος εκπρόσωπός της που θα ήθελε να σχολιάσει. Να κάνω και εγώ δύο παρατηρήσεις λοιπόν. Πρώτον, μια διευκρίνηση. Εκτίμησα αυτά που είπατε κυρία Μπίλτερ, όμω μια παρατήρηση. Το Erasmus Plus και η Δημιουργική Ευρώπη έχουν ω νομική βάση ε, τέτοια διάταξη που επιτρέπει τη συνεργασία με τρίτε χώρε. Το Erasmus Plus ε, ε, σχετίζεται με δύο γραμμέ, Πρώτα απ' όλα το Comenius που έχει να κάνει με σημαντικότατες μορφές συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή σχολικών ιδρυμάτων με διάφορους τρόπους και διαφόρων χωρών αλλά και την ανάκτηση των απαραίτητων αρμοδιοτήτων για την ε, ε, αναπαλαίωση ή την συντήρηση σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς. Αλλά και το Εράσμος Μούντου, τα πλαίσια του έρασμου είναι μια υπηρεσία εθελοντική στην ε, Ευρώπη που πολλέ φορέ λαμβάνει σαρκά και ουσιαστά και σε τρίτες χώρες. Νομίζω ότι ο κύριος Σφέγκερ θα είναι ο ε, μόνιμος συγκεκριτής για τα θέματα του Erasmus Plus. Για τη δημιουργική Ευρώπη κατά τα άλλα, η έκκλησή μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εξή, διότι ανησυχούμε λίγο Προβλέποντα τα πλαίσια τη Δημοτικής Ευρώπη ε, δημιουργήσει ε, συμφωνίε με τρίτε χώρε για να ευνοηθεί η συνεργασία σε πολιτιστικό επίπεδο στην, στον τομέα της δημιουργίας. Όμως προς στιγμή οι συμφωνίε έχουν γίνει με κάποιε χώρε τη Ανατολική Ευρώπη Ευρώπης και όχι τη Μεσογείου, του Νότου. Η την Ισία είναι ένα καλό παράδειγμα. Θέλουμε λοιπόν να παρατρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει κίνητρα για να συναθούν περισσότερε τέτοιε συμφωνίε. Και χρειάζονται και πρόσθετα τα κονδύλια. Πρέπει και αυτό να το εξολογήσουμε, διότι σε φτωχότερε χώρε κάποιε φορέ οι συνεισφορέ μα είναι μόνο συμβολικέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να προσθέσει κάτι. Εάν όχι, να προχωρήσουμε. Μάλλον όχι, οπότε στη φάση αυτή να θυμίσω σε όλου ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 21 Μαρτίου και να ευχηθώ καλή δουλειά στο συνάδελφο Ζαμπάσκη. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο το οποίο μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό και μας ενδιαφέρει, να ευχαριστήσω για την παρουσία τους τον Διευθυντή της Γενικής ε, Διεύθυνσης Τζαντιέρη και τους δύο προσώπους της Eurostat για την πολιτιστική στατιστική τον ε, δόκτορα Μέρση και την κυρία Ντονσάσκαν Σάσκαν σωστά διαβάζω το όνομά και μετά την εμπειρογνώμονα της ΣΥΑ η οποία θα μας μιλήσει για διάφορες πολιτικές διαστάσεις του οπτικοακουστικού κλάδου. Να θυμίσω απλώς ότι η μέλη... Παρακαλώ καθίστε. παρακαλώ πάρτε θέση. να θυμίσω Prego, Valentina Montalto. Volevo solo ricordare... Eh, να θυμίσω απλώς ένα πράγμα προκαταρτικά. Όπως τα γνωρίζετε, στο άρθρο 15 του Κανονισμού για τη Δημιουργική Ευρώπη, το Κοινοβούλιο εξέφρασε μια συγκεκριμένη απέτηση. Η Επιτροπή να διεξαγάγει μια μελέτη εντεκτύπου για να δει κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε δεδομένα στον τομέα του δημιουργικού κλάδου και όχι μόνο στον οπτικό ακουστικό όπου υπάρχει ένα καταπληκτικό παρατηρητήριο στο Στρασβούργο και να παρουσιάσει τα πορίσματα και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Έχετε λοιπόν το έγγραφο και θέλω να θυμίσω δύο πράγματα για το θέμα. Ότι έχουμε 20 χρόνια από τότε που τοποθετήθηκε το Συμβούλιο των Υπουργών, νομίζω το 94-95, και μίλησε για την ε, ανάλυση και την εμβάθυνση στα στατιστικά στοιχεία στον πολιτιστικό κλάδο. Στρατηγική σημασία για να καταλάβουμε και τον αντίκτυπο των πολιτικών και την συνεισφορά των τομέων αυτών στην ανάπτυξη και την ανάληψη αρμοδιοτήτων αλλά και την οικονομία. Επίσης είναι σημαντικό ε, ότι από το 2012 η Eurostat δημιούργησε μια ειδική μεθοδολογία την οποία μοιράζεται με την ΕΣΝΕΤ και χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά, τα συμπεριλαμβάνει στις μελέτες της ε, ανακράτως. Αυτό έγινε ένα στοιχείο που έλαβε υπόψη του σοβαρά και ο ΑΣΕ, οπότε τα στατιστικά στοιχεία για την ε, πολιτιστική παραγωγή και τη δημιουργία αποτελούν μέρος του δίκτυ για την ε, ευημερία, όχι δηλαδή να τα υπολογίζουμε όλα βάσει του ΑΕΠ. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά που κάνει σε αυτό το επίπεδο η Eurostat και είναι πραγματικά ε, έντονη η επιστημονική συνεργασία εδώ αλλά πραγματικά θέλουμε να θυμίσουμε και αυτή τη σαφή ένδειξη με το πράσινο βιβλίο για τη Δημιουργική Ευρώπη και μιλώντας για τον πλέον κατάλληλο τομέα που ανοίγει δρόμους για τις απαιτήσεις που δημιουργούνται και ως προς τους πόρους και ως προς τη χρηματοδότηση είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σύνολο δεκτών συγκρισίμων οι οποίοι να είναι και καταλληλότεροι και ευστοχότεροι και να καλύψουν την πολιτιστική μέρημνα της Ευρώπης όπως έχει δημιουργηθεί. Φαίνεται να είμαστε κάπως ε, ε αμελείς σε ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό όπως η Ευρώπη του πολιτισμού σε καιρούς κρίσης. Ε, να σας δώσω λοιπόν το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και παίρνετε το μικρόφωνο. Uh, so, thank you very much, Madam Chair. ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το έργο μας ε, για τα στατιστικά στοιχεία για τον πολιτισμό στο Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό για σας και για την βοήθεια που έχει δοθεί. Σας ευχαριστούμε. Ήταν πολύ σημαντικό και για τα κράτη-μέλη. Είναι προτεραιότητα στο έργο μας με τα κράτη-μέλη να υπάρξει ο συντονισμό για το θεματολόγιο το ευρωπαϊκό για τον πολιτισμό και σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εντάσσεται απόλυτα στις προτεραιότητες για ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης του Γιούγκερ. Πρέπει να καταδείξουμε τις επιπτώσεις στον τομέα του πολιτισμού υπέρ της Ευρώπης για την οικονομία και την κοινωνία. Έχουμε δύο παρουσιάσεις με τους συναδέλφους της Eurostat και με την, ε, τους υπεύθυνους για την feasibility study, τη μελέτη εφικτότητας. Είμαστε ικανοποιημένοι και ιδιαίτερα ευχαριστημένοι για την δυνατότητα οι συνάδελφοι της Eurostat να είναι παρόντες. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα δώσω αμέσω ε, τον λόγο. Χαιρόμαστε υπό την δημιουργικότητα στην Ευρώπη να καλύπτουμε αυτό το έργο για να μπορέσουμε στον τομέα της υποστήριξης που πρέπει να δοθεί για καλύτερες πολιτικές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη και για να υποστηριχθεί και το έργο του Κοινοβουλίου εξάλλου. Θα δώσω τώρα τον λόγο πρώτα, κυρία Πρόεδρε, στους συναδέφους της Eurostat, αν επιτρέπετε. Ευχαριστώ. Εργάζομαι στη Eurostat είναι μια γενική διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η δική μας και σας ευχαριστούμε που μας προσκαλέσατε και μας φιλοξενείτε σήμερα και μετά το επίπεδο προσδοκιών που παρουσιάστηκε από την Πρόεδρο και τον συνάδελφο ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να σας δώσουμε κάποια ικανοποιητικά στοιχεία διότι οι προσδοκίες σας είναι πάρα πολύ υψηλέ βέβαια. Τώρα με στατιστικά στοιχεία, όταν έχει κανείς στατιστικά στοιχεία μπροστά του, το πρώτο που πρέπει να βρούμε είναι τι εννοούμε με τον πολιτισμό και τα στατιστικά στοιχεία για τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός έχει πολλές έννοιες και σημασίες και πολλές αναφορές και γι' αυτό οι στατιστικές δραστηριότητες για να μπορέσουμε να έχουμε στοιχεία για αυτό το περίπλοκο θέμα προτεραιότητα είναι να τραβήξουμε τις διαχωριστικές γραμμές. Ποιο είναι το πεδίο για το οποίο κάνουμε λόγο και πρέπει να μετρηθεί και τι μπορεί να μετρηθεί υπό το πρίσμα των στατιστικών στοιχείων. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε επί παντός του επιστητού όλα τα μετρήσιμα στοιχεία, αλλά τα ουσιοδέστερα για αυτό το πεδίο πρέπει να μπορέσουμε να τα καλύψουμε. Κάνοντας αυτό εκπονήσαμε όπως αναφέρθηκε από την Πρόεδρο, ένα πλαίσιο πλαίσιο που καθορίζει και εντοπίζει παιδεία που είναι τα παιδεία των πολιτιστικών δραστηριοτήτων όπως πολιτισμός, παράδοση, τέχνες, αποκινούμε τις λειτουργίες. Λειτουργίες για την δημιουργία παραγωγή πολιτισμικών και πολιτιστικών προϊόντων, στην παιδεία, εκπαίδευση, δημιουργικότητα και την διαχείρισή τους. Έχουμε πολιτισμικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που προσπαθούμε να περιγράψουμε με αυτά τα στοιχεία από πλευράς μας στο έργο μας. Λοιπόν, τι εκπονήσαμε σε αυτό το πλαίσιο όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία αυτή τη στιγμή. Είναι ακόμα σε εμβρική μορφή, ε, ε, αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε Έχουμε στοιχεία για την απασχόληση στο, πεδίο του πολιτισμού και την οικονομική πτυχή όσον αφορά τα πολιτισμικά θέματα. Στοιχεία επίσης ε, του διεθνούς ε, εμπορίου όσον αφορά υπηρεσίες και αγαθά. Συμμετοχή στον πολιτισμό, δηλαδή την κατανάλωση εντό εισαγωγικών πολιτισμικών προϊόντων και δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον ρόλο των νέων τεχνολογιών μέσα στο πλαίσιο της διάχυσης ε, και διάδοσης προϊόντων και κατανάλωσής τους και όσον αφορά και τις δαπάνες για τα αγαθά και τις υπηρεσίες υπηρεσίες ε, ποιες είναι αυτές. Αν το πάρουμε ένα, τα πάρουμε ένα-ένα, βήμα προς βήμα και για την απασχόληση, γιατί επ' αυτής έχουμε μάλλον τα καλύτερα, πιο αξιόπιστα στοιχεία αυτή τη στιγμή διαθέσιμα, μπορείτε να δείτε ίσως αν έχετε μπορείτε να δείτε και ε, αρκετά μακριά αυτό το γράφημα με τις ε, με τα στοιχεία που αναφέρονται λυπούμε αν δεν είναι πάρα πολύ ευδιάκριτα τέλος πάντων Εντάξει. Βλέπετε ότι η απασχόληση στον πολιτισμό το 2014 είναι 2,9% της συνολικής απασχόλησης στην Ευρώπη. 2,9% μπορεί να θεωρηθεί μεγάλο ποσοστό ή και χαμηλό, μικρό μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει εδώ και μία ας το πω έτσι ε, τομή όσον αφορά τις ε, έρευνες ε, για αυτό το χρονικό διάστημα. Για να σας δώσω το μέγεθος, η απασχόληση στον πολιτισμό είναι περίπου του ιδίου επίπεδου όπως στην ενημέρωση και πληροφόρηση των τομέα ICT και των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής περίπου ο ίδιος ε, αριθμός απασχολούμενων όπως επίσης και στις, ασφάλειες, στις ασφαλιστικές εταιρείες και στις ε, τραπεζικές δραστηριότητες. Τρία περίπου τους εκατό εκεί είναι πολύ ε, περισσότερο θα λέγαμε σε σχέση για παράδειγμα ε, όσον αφορά τα στοιχεία για την ε, ενέργεια. Αυτά τα στοιχεία σας δίνουν κάποιες πληροφορίες, κάποια μεγέθη. Αυτά μπορούν να συγκριθούν με την εξέλιξη των στοιχείων απασχόλησης πάνω πάνω στο γράφημα. Έχετε την εξέλιξη της απασχόλησης στην Ευρώπη μέχρι το 2014 και βλέπετε λόγω της κρίσης υπήρξε φθήνουσα πορεία, μείωση της απασχόλησης στην Ευρώπη κατά το διάστημα αυτό, όμως ο πολιτισμικός τομέας ήταν ανθεκτικός, άντεξε, δεν υπέστη εκείνος τις, επι, τις επιπτώσεις της κρίσης όσον αφορά την απασχόληση και έτσι δεν υπήρξε τέτοια φθήνουσα πορεία σε αυτόν. Αυτά για την απασχόληση. Πρέπει να υποφεληθούμε του γεγονότος ότι στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα έχουμε τεράστιες βάσεις δεδομένων και στοιχείων και μπορεί κανείς να δει τα στοιχεία για την απασχόληση σε σύγκριση και με άλλα στοιχεία που είναι διαθέσιμα και που περιγράφουν εκείνα τις υπόλοιπες δραστηριότητες του οικονομικού τομέα ή άλλων τομέων. Εδώ για παράδειγμα αναχώρα έχουμε τη διασύνδεση στον αριστερό άξονα το ΑΕΠ ανακεφαλήν και κάτω στην κάτω πλευρά την πολιτισμική απασχόληση. Δεν θα ισχυριστώ ότι δεν υπάρχει κάποια διασύνδεση. Όχι. Αφήνω σε εσά να ανοιχνεύσετε την διασύνδεση αυτή. Δεν είναι δική μας δουλειά να αναλύσουμε υπερβολικά αυτά τα στοιχεία. Μπορείτε όμως να δείτε ότι υπάρχει μια διασύνδεση. Μπορεί κανείς να το δει αυτό. Σε σχέση με την αναλογικότητα, την αναλογία, όχι τον αριθμό ατόμων ως απόλυτο μέγεθος, αλλά την επίπτωση αυτή όσον αφορά τον τομέα της, ε, του πολιτισμού και το ΑΕΠ ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, ιδιομορφίες ε, που έχουμε σε σχέση με το Λουξεμβούργο. Μπορεί κανείς να δει τα άλλα όμως στοιχεία στο γράφημα αυτό που δίνουν κάποια στοιχεία για την οικονομική, την οικονομική αξία των πολιτιστικών δραστηριοτήτων η πρόεδρος είχε την ευμένεια να μιλήσει για την ε, ε, ποιότητα ζωής και την ευημερία. Στο ίδιο ε, επίπεδο αυτό, υποκειμενική ποιότητα ζωής και απασχόληση στον τομέα του πολιτισμού. Μπορεί κανείς να δει τη διασύνδεση μεταξύ της ποιότητας διαβίωσης, όπως υποκειμενικά την μετρούν και την αισθάνονται οι πολίτες, και την απασχόληση, την, τον άξονα ή το συσχετισμό με την απασχόληση. Και πάλι αυτό δεν είναι πρόβλημα της Eurostat. Παράγουμε εμείς αυτά τα στοιχεία και αφήνουμε την ανάλυση στους αρμοδίους, τους εμπλεκόμενους που έχουν το καθήκον και την ίσως ευχαρίστηση κιόλας να τα αναλύουν για να δουν τις επιπτώσεις τους πάλι στο επίπεδο της απασχόλησης. Οι οικιανοί στιγμοί, οι τελίτσες οι μπλε σας δείχνουν αναχώρα την αναλογία του τριτογενούς πεδίου ε, των ε, ανθρώπων που είναι ε, καταρτισμένοι σε αυτό το πεδίο, σε αυτό το επίπεδο. Αριστερά βλέπετε στην αριστερή πλευρά 32% περίπου των απασχολούμενων στον τομέα αυτό έχουν ένα πτυχίο του, ε, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τώρα με τον κίτρινο άξονα βλέπετε ότι η αναλογία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην απασχόληση στον πολιτισμικό τομέα είναι πολύ υψηλότερη η αναλογία αυτή. Όχι μόνο έχουμε 2-3% της απασχόλησης λοιπόν των ατόμων που εργάζονται στον πολιτισμό, συνολικά, αλλά βλέπουμε επίσης ότι αυτές οι θέσεις απασχόλησης είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένες με πολύ προηγμένα προσόντα θα έλεγα όσον αφορά τις ε, δεξιότητες και ικανότητες των εργαζομένων. Όταν κάνουμε λόγο τώρα για αυτές τις ε, πρωτοβουλίες ε, σε αυτόν τον τομέα, στον οικονομικό τομέα κυρίως για τον πολιτισμό, αυτό που βλέπουμε σε αυτό το γράφημα είναι ότι περίπου 5% της πρόσθετης αξίας, 5% στις της πρόσθετης αξίας 5% στις υπηρεσίες, στον τομέα των υπηρεσιών, οφείλεται το 5% σε πολιτισμικές δραστηριότητες. Πάλι αυτό μπορεί να φανεί σε κάποιο μικρό ποσοστό, όμως από την άλλη πλευρά 5% συνολικά της πρόσθετης αξίας ε, που δημιουργείται και παράγεται είναι ένα αξιόλογο ποσοστό και μπορεί να δει κανείς ότι υπάρχουν και μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά το μερίδιο αυτών των πολιτιστικών πολιτικών δραστηριοτήτων στον τομέα των υπηρεσιών, στον πολιτισμό. Μπορούμε επίσης να δούμε και κάτι άλλο. Ποιοι είναι ποιε είναι αυτέ οι επιχειρήσει και πρωτοβουλίε δραστηριότητε που παρέχουν, δημιουργούν αυτή την πρόσθετη αξία. Είναι τηλεοπτικέ εκπομπέ, ραδιοφωνικέ εκπομπέ, ταινίε, ε, στην τηλεόραση διάφορες ε, δραστηριότητε, εφημερίδε, δημοσιεύματα, περιοδικά και άλλα δημοσιεύματα, άλλε δραστηριότητε στον τύπο. Μπορούμε λοιπόν να δούμε τώρα και αυτό το γράφημα και αυτό αυτά τα στοιχεία μέσα στο πλαίσιο των στοιχείων που παρέχονται από την Ευρωστάτ. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που μπορούμε να προσφέρουμε είναι το τμήμα του διεθνούς εμπορίου, του παγκόσμιου εμπορίου όσον αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Εντοπίζοντας και ε, ταυτοποιώντας στο διεθνές εμπόριο ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά τα προϊόντα στον πολιτισμικό τομέα που δημιουργούν αυτή την πρόσθετη αξία. Εισαγωγές και εξαγωγές. Βλέπει κανείς ότι διακυμαίνονται. Υπάρχει μια διακύμανση ανά έτος. Δεν είναι εύκολο να βρει κανείς τα πρότυπα αυτής της εξέλιξης. Όμως υπάρχουν τα στοιχεία και η κλίμακα όσον αφορά τα δισεκατομμύρια ευρώ στα οποία μετρούμε αυτά τα στοιχεία ε, στην κλίμακα αυτή. Δηλαδή εδώ δεν έχουμε μόνο χιλιάδες ή εκατομμύρια αλλά δισεκατομμύρια ευρώ όσον αφορά αυτές τις εξαγωγικές ή εισαγωγικές δραστηριότητες. Περί τίνος πρόκειται σε αυτά τα αγαθά. Πρόκειται κυρίως για έργα τέχνης, βιβλία, αντίκες, ε, ε, αγαθά στον τομέα αυτών. Με ποιους εμπορευόμαστε αυτά τα αγαθά. Μια άλλη ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εξάγουμε λοιπόν προς τις ΗΠΑ, στην Ελβετία, προς την Ελβετία το Χονγκ Κόνγκ και εισάγουμε από την Κίνα, ΗΠΑ και Ελβετία. Τώρα, αυτό που εισάγουμε, αυτά που εισάγουμε από την Κίνα, ίσως θα σας φανεί περίεργο, αξιοπερίεργο, αλλά είναι κυρίω, κυρίως <clears throat> χειροποίητα ή μεταποιημένα αγαθά που αφορούν ε, ηλεκτρονικά παιχνίδια, ε, περιεχόμενο ηλεκτρονικών και ε, τηλεοπτικών παιχνιδιών, βλέπουμε εδώ σε σχέση με το σχέδιο και το περιεχόμενο δεν προέρχονται, δεν είναι δημιουργήματα των ίδιων των Κινέζων, προϊόντα των ίδιων των Κινέζων, αλλά παράγονται στην Κίνα. Τώρα, συμμετοχή. Με ποιο τρόπο συμμετέχουν οι Ευρωπαίοι, η Ευρώπη συνολικά στα πολιτιστικά θέματα. Έχουμε κάποια στοιχεία πληροφοριακά. Θα σας δώσω, θα σας δώσω κάποια στοιχεία σε σχέση με αυτά που έχουμε συλλέξει εδώ. Για παράδειγμα, έχουμε το ποσοστό του πληθυσμού που έχει διαβάσει πάνω από 10 βιβλία το, προηγούμενο έτος, 12 μήνες. Και αναφύλλω, άνδρες, γυναίκες. Το μπλε οι άνδρες, ε, το κίτρινο οι γυναίκες. Οι γυναίκες είναι πολύ πιο πάνω λοιπόν κυρίες και κύριοι. Θα μπορούσαν οι άνδρες να είχαν καλύτερες επιδόσεις. Θα μπορούσαν οι επιδόσεις τους να είναι καλύτερες. Μπορούμε επίσης να ρίξουμε μια ματιά και να δούμε ποια είναι η συχνότητα, πόσο συχνά πάνε σε ε, συναυλίες, ε, στο θέατρο. Και εδώ ίσως θα είναι ενδιαφέρον. Πρέπει να είναι ενδιαφέρον να δει κανεί το ποσοστό εκείνων που δεν πάνε ποτέ σε συναυλίες, κονσέρτα, σε θεατρικές παραστάσεις ε, σε σχέση με το γράφημα που μπορεί να το δει κανείς ε, για αυτό το ποσοστό και μπορεί να φτάνει κανείς ε, πολλές φορές και σε πάρα πολύ ψηλό ποσοστό αυτό το μερίδιο του πληθυσμού. Ένα άλλο παράδειγμα. Επισκέψεις ε, μουσείων, εκθέσεων ε, ε, όσον αφορά τις πολιτιστικές, πολιτισμικές εκθέσεις περιεχομένου πολιτισμικού οι επισκέψεις αυτές είναι πολύ σημαντικές για εκείνους που έχουν ανώτερη εκπαίδευση και είναι πολύ μικρότερη σημασία για εκείνους που έχουν χαμηλότερο επίπεδο παιδείας και εκπαίδευσης πράγμα το οποίο συναρτάται φυσικά με την, ε, τις επιδόσεις αυτές και την παιδεία των ατόμων τέτοιου είδου ε, δραστηριότητες που μπορεί κανείς να τις ε, έχει υπόψη του που μπορούν με αυτόν τον τρόπο να εξηγούνται. Επίσης τώρα σε σχέση με την, το ITC για πολιτισμικές δραστηριότητες αποϊλοποιημένη ας το πούμε έτσι ε, δραστηριότητα τι γίνεται στο ηλεκτρονικό επίπεδο στο διαδίκτυο τι, ποιες δραστηριότητες ε, ακολουθούνται και εδώ βλέπουμε ότι η χρήση του διαδικτύου για πολιτισμικές δραστηριότητες ηλικία στην κάτω πλευρά βλέπετε την αύξουσα ε, πορεία σε σχέση με την ηλικία των ατόμων. Όσο νεότεροι είναι τόσο περισσότερη δραστηριότητα και στη νεότερη κατηγορία 16 24 ετών το, τα παιχνίδια έχουν πριν τα ανέβω κυρίαρχο ρόλο. Ωστόσο 65% των νέων από 16 έως 24 ετών χρησιμοποιούν το διαδίκτυο το χρησιμοποιούν για να συμβουλευτούν, να χρησιμοποιήσουν ε, τις ε, ιστοσελίδες ε, εφημερίδων, περιοδικών. Μπορεί κανείς φυσικά να διασκεδάζει συλλέγοντας τέτοια τέτοιες πληροφορίες και τέτοια στοιχεία όσον αφορά τις ειδήσει, δημοσιεύματα, εφημερίδες από ιστοσελίδες. Η αγορά βιβλίων στο διαδίκτυο έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία. Εδώ βλέπουμε τη σύγκριση 2009-2015. Μουσική, περιοδικά, <clears throat> εισιτήρια. Δεν είναι ακόμα η κυριότερη δραστηριότητα στο διαδίκτυο ακόμα αυτή. Ωστόσο, οι αγορές αυτές προοδεύουν, αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου και έχοντας και μία προσέγγιση όσον αφορά τα νοικοκυριά και τις δραστηριότητες τους, τις διαφορετικές οικογένειες, ποια είναι η κατανάλωση, ποια είναι η δαπάνη στα νοικοκυριά για αυτές τις υπηρεσίες και αγαθά. Έχουμε κάποια στοιχεία και για αυτό επίσης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην ΕΕ τα νοικοκυριά πάνω από 3% του, των εσόδων τους, του εισοδήματός τους ε, το καταναλώνουν, το αναλώνουν για την αγορά τέτοιων αγαθών και υπηρεσιών. Σας υπενθυμίζω ότι περίπου 60%, 60 του συνόλου των δαπανών δαπανώνται σε τρεις άξονες στέγαση, διατροφή, μεταφορές και το υπόλοιπο 40% ε, στη διακριτική ευχαίρεια της κάθε οικογένειας είναι το πώς θα δαπανηθεί για να υπάρχει κάποια συγκρισιμότητα όσον αφορά την ε, δαπάνη ας πούμε για την υγεία περίπου του ιδίου ύψους του ιδίου επίπεδου 3,5% και το ίμιση όσον αφορά τις ε, δραστηριότητες αναψυχής και διασκέδασης και πολύ περισσότερο σε σχέση με τη δαπάνη για ε, τον καπνό και τα ινοπνευματόδη. Τώρα, τι συνεπάγονται όλα αυτά, τι αγοράζουν με όλα αυτά τα νοικοκυριά συνδρομές ε, όσον αφορά τηλεοπτικές εκπομπές, ραδιοφωνικές εκπομπές περιοδικά, ε, συσκευές τηλεόρασης πηγαίνουν στον κινηματογράφο, στο θέατρο και όλες τις άλλες ε, συναφείς δραστηριότητες τιμές και οι τιμές είναι αρκετά ενδιαφέρουσες ως στοιχείο για τις δραστηριότητες τον τομέα των προϊόντων και υπηρεσιών. Εδώ έχουμε την εξέλιξη των τιμών για αυτά τα προϊόντα στην ε, πάροδο των ετών. Μπορεί κανείς να δει εδώ ότι υπάρχει μία μείωση σε σχέση με τις τιμές όσον αφορά το hardware δηλαδή τις συσκευές τηλεόρασης, ε, ε, τις, τις τηλεοράσεις, τις συσκευές ηλεκτρονικών υπολογιστών λοιπά. Μείωση τιμών σε σχέση με την περίοδο αυτή είναι οι τιμές για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις συσκευές ε, τηλεοπτικές και τα λοιπά μειώνονται και με την πράσινη γραμμή με την εξαίρεση που μπορεί κανείς να δει εδώ σε σχέση με το στοιχείο της μείωσης των τιμών μπορεί κανείς ε, να δει ιδιαίτερα σε σχέση με την ε, διασύνδεση στο διαδίκτυο και την ελεύθερη πρόσβαση σε ταινίες και μουσικά προϊόντα και μουσική. Για να ολοκληρώσω θα μπορούσα να σας δείξω μια ολόκληρη σειρά στοιχεία, κάποια στοιχεία. Είναι στοιχεία τα οποία παράγουμε για το, τις δαπάνες μας. Το ενδιαφέρον με την χρήση των στατιστικών στοιχείων της Eurostat έγκυται στο ότι τα εναρμονισμένα αυτά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών χωρών και των δραστηριοτήτων τους με μεγάλη αξιοπιστία και συνδέονται και με άλλα στοιχεία ε, τα οποία παράγονται. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα και τη Eurostat υπάρχει συγκεκριμένο όφελος διότι υπάρχει πρόσθετη αξία διότι μπορούν να συγκριθούν αυτά με άλλα στοιχεία του συστήματος ε, όσον αφορά για παράδειγμα το ΑΕΠ και την ποιότητα ζωής και διαβίωσης. Έχουμε εκπονήσει διαφορετικές προσεγγίσεις, απασχόληση, συμμετοχή στο εμπόριο και προσέγγιση όσον αφορά αυτά τα στοιχεία. Θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτά τα στοιχεία ε, επί τακτής, τακτής βάσεως ε, ε, συλλέγονται. Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι προέρχονται από διαφορετικές υφιστάμενες διαθέσιμες πηγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα στοιχεία. Δεν υπάρχει μια ειδική συλλογή στοιχείων που να αφορά τον τομέα του πολιτισμού αυτή τη στιγμή, μέχρι σήμερα δηλαδή. Είναι κάποια από αυτά τα στοιχεία ετήσιας βάσης, ε, συλλογές επί ετήσιας βάσης. Άλλα είναι με πολιετής, ε, με βάσης δεδομένων που είναι στη διάθεσή μας. Θα μπορούσε κάποια ταξινόμηση στατιστική σε αυτό το πεδίο να πει κανείς ότι δεν είναι αρκετά αξιόπιστη ώστε να απεικονίζεται με κάθε σαφήνεια ο τομέας του πολιτισμού. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να δώσουμε συνέχεια και να μην εμείνουμε σε αυτό, σε αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει λοιπόν εδώ η θετική αυτή πτυχή και πρέπει να συνεχίσουμε ώστε να βελτιωθούμε περισσότερο και να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες επιδόσεις διότι όλο και περισσότερο τα πολιτισμικά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Τι σημαίνουν όλα αυτά Μπορείτε ήδη να το δείτε στην ιστοσελίδα της Eurostat βέβαια, αλλά είναι σε επέκταση, επεκτείνεται ο τομέας και τα στοιχεία και οι στατιστικές αναλύσεις θα ακολουθήσουν και θα, υπάρξουν, θα υπάρξει παραγωγή στοιχείων για να καλυφθούν αυτές οι δραστηριότητες εντός ολίγου και εμείς προβλέπουμε ότι θα υπάρξει διεύρυνση και επέκταση αυτών των ε, στοιχείων και πηγών. Προσπαθούμε να καλύψουμε με καλύτερο τρόπο τις ε, πολιτισμικές δραστηριότητες και τη συλλογή αυτών των στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά υπάρχουν πράγματα τα οποία βρίσκονται υπό εξέλιξη και πρέπει να μπορέσουν να προαχθούν η ταξινόμηση είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί. Παρακολουθούμε τα θέματα ταξινόμησης και ονοματολογίας σε παγκόσμια κλίμακα. Μπορεί να φαίνεται απλό αυτό, αλλά είναι τόσα πολλά και διαφορετικά τα θέματα και οι, πρωτο, προτεραιότητες και πρωτοβουλίες για την ταξινόμηση που δεν είναι πολύ εύκολο να αγνοήσει κανείς ή να μην λάβει υπόψη ότι κάποιοι τομείς έχουν καλύτερη παρουσίαση από άλλους. Αυτά από πλευρά μου σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Δεν τελειώνει. Βρίσκεται υπό εξέλιξη ρευστό αυτή η διαδικασία. Δεν τελείωσε. Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η εξήγησή σας για την πολύ σημαντική δουλειά που κάνετε. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Τερέσα Μοντάλτο. Να πω πως θα δημοσιευθεί το επόμενο survey τον Ιούνιο του 2016 και βεβαίως θα μοιραστεί σε όλους τους συναδέλφους. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη συνεισφορά ε, την οποία θα πρέπει να δούμε ε, προσεκτικά. Τα ε, έγγραφα ακόμα δεν έχουμε μπορέσει να σας τα μοιράσουμε αλλά σίγουρα, σίγουρα μετά τη συνεδρία θα τα έχετε. Παρακαλώ πολύ Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να παρουσιάσετε το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει γίνει η δουλειά σας. Και σας ευχαριστώ πολύ ε, που βοηθήσετε και εσείς στην οργάνωση της σημερινής συνάντησης. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας. Είναι τιμή για μένα να είμαι εδώ. Θα σας παρουσιάσω τα βασικά ευρήματα, συμπεράσματα και συστάσεις για τη μελέτη αυτή, η οποία έγινε όπως υπόθηκε στα πλαίσια αυτής της κοινή προσπάθειας να βελτιωθούν τα στατιστικά στοιχεία για τον πολιτισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πω δύο λόγια για το KEA που είναι ένα ερευνητικό κέντρο με βάση στις Βρυξέλλες εξειδικευμένο στον δημιουργικό και στον πολιτιστικό κλάδο. Εμείς έχουμε προετοιμάσει επίσης και δύο εκθέσεις που έγιναν και πάλι με προτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 6 και το 9 η οικονομία του πολιτισμού στην Ευρώπη είναι η πρώτη χαρτογράφηση που έγινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτού του κλάδου και μετά είχαμε και τις επιπτώσεις του πολιτισμού και της δημιουργικότητας ως όχημα ε, για την καινοτομία κάτι το οποίο ε, γράψαμε, συντάξαμε το 2009 που ήταν το έτος δημιουργικότητας. Έχουμε λοιπόν και τις κατοπινές μας έρευνες στον ε, συγκεκριμένο χώρο για να ευαισθητοποιήσουμε και να μάθουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις ευρείας κλίμακας του κλάδου αυτού στην ευρωπαϊκή κοινωνία ευρύτερα. Όπως υπόθηκε στην αρχή της σημερινής συνεδρίασης, το βασικό θέμα είναι το πώς μπορούμε να μετρήσουμε αυτές τις επιπτώσεις, τον αντίκτυπο που έχει. Όπως είπε και η κυρία Κώστα, έχουν συμβεί πάρα πολλά τα τελευταία 20 χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξεκινήσαμε το 1995 με την υιοθέτηση του πρώτου ψηφίσματος για την βελτίωση των πολιτιστικών στατιστικών προς την οικονομική ανάπτυξη και μετά στήθηκε μια τεχνική ομάδα εργασίας που είχε ως σκοπό να βελτιώσει τις μεθοδολογίες συλλογής δεδομένων για τον κλάδο. Η Eurostat λοιπόν κάνει αυτή την προσπάθεια την οποία μόλις σας παρουσίασα και για να συμπληρώσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό το φιλόδοξο σχέδιο ο κανονισμός που έστησε το πρόγραμμα Creative Europe ε, προέβλεπε και μία μελέτη σκοπιμότητας έτσι ώστε να εξερευνηθούν κάποιοι νέοι μηχανισμοί συλλογής δεδομένων για να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμα νέες μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης στατιστικών δεδομένων στον κλάδο αφήνοντας εκτός τον κλάδο του όπτιο ακουστικού γιατί εκεί έχουμε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο που κάνει πολλή δουλειά, ε, ποιοτική δουλειά και λεπτομερή δουλειά. Ακολουθήσαμε λοιπόν την εξής μεθοδολογία. Πρώτα απ' όλα συνεργαστήκαμε πολύ στενά με τη Eurostat η οποία μας έστειλε πολύ σημαντικά έγγραφα για να μπορέσουμε εμείς καταρχήν να περάσουμε ε, ε, μια πρώτη ματιά της επίσημες στατιστικές και να δούμε τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει, ποια κενά πρέπει να αντιμετωπίσουμε και μετά, και αυτή είναι η προσθέμενη αξία της δουλειάς μας, χαρτογραφήσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενδεχόμενες εναλλακτικές πηγές που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να έχουμε μια ευρύτερη κατανόηση του κλάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διοικητικά αρχεία, ε, big data ε, που βρίσκονται online, όπως επίσης πολιτιστικά παρατηρητήρια και αξιολογήσαμε τα κενά που υπάρχουν μεταξύ επισήμων στατιστικών στοιχείων και εναλλακτικών πηγών, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε κάποιες βασικές συστάσεις και σενάρια εφαρμογής αυτών. Τι διαπιστώσαμε. Υπάρχει μια σειρά ζητημάτων και προκλήσεων που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν εδώ στο συγκεκριμένο χώρο. Προκλήσεις που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένους κλάδους και κάποιες άλλες που είναι περισσότερο εγκάρσιες και καλύπτουν όλο τον κλάδο τον πολιτιστικό δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για όλα. Θα πω όμως δύο λόγια για το Διεθνές Σύστημα Ταξινόμησης, για παράδειγμα. Οι διάφοροι κωδικοί μέσω των οποίων η οικονομική δραστηριότητα και η απασχόληση και οι θέσει εργασία ε, αναγνωρίζονται, δεν είναι απολύτω προσαρμοσμένε στο να κατανοήσουν τι γίνεται στο δικό μα κλάδο. Γιατί κάποιε δραστηριότητε είναι δύσκολο να απομονωθούν και να εντοπισθούν ως πολιτιστική δραστηριότητα. Και αυτό αληθεύει κυρίω για τα παιχνίδια βίντεο, ε, για τη μουσική κτλ. Και υπάρχουν και κάποιοι κλάδοι που καλύπτονται λιγότερο από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δηλαδή είναι ε, φεστιβάλ, ε, κάποιες ε, βιβλιοθήκες πολιτιστικές, πολιτιστικής κληρονομιάς, κάποια τα οποία καλύπτουν διάφορους χώρους που είναι για παράδειγμα ο σχεδιασμός και η παραγωγή παιχνιδιών Και το βασικό είναι ότι ο χώρος αυτός ε, αποτελείται από μια πολύ μεγάλη γκάμα μικρών και πάρα πολύ μικρών επιχειρήσεων και είναι δύσκολο να παρακολουθήσουμε την εξέλιξή τους σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Ξέρουμε πως υπάρχουν στοιχεία, αλλά δεν παρουσιάζονται αυτά πάντα ψηφιακά και πολλές φορές δεν έχουμε και στοιχεία για την εμπορία των πολιτιστικών αγαθών όπου ε, σε περίπτωση που έχουμε άλλα στοιχεία, όπως για παράδειγμα τα ηλεκτρονικά βιβλία ή ανταλλαγή υπηρεσιών, όπου έχουμε δηλαδή μια ε, εξαήλωση των αγαθών που ανταλλάσσουμε, είναι πλουθήσουμε ε, τις εξελίξεις. Οι εναλλακτικέ πηγές λοιπόν πώς μπορούν να μας βοηθήσουν. Με τρεις τρόπους. και να συμπληρώσουν τις πληροφορίες που έχουμε ε, και οι οποίες ε, παρέχονται από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Καταρχήν συμπληρώνουμε τεκμήρια και στοιχεία για κλάδους που δεν καλύπτονται τόσο πολύ ε, από τα επίσημα ευρωπαϊκά. Για παράδειγμα, βιβλιοθήκες, το έγμους μπορεί να μας δώσει κάποια στοιχεία. Το έγκυτα, με συγχωρείτε. Και έχουμε και κάποια φαινόμενα τα οποία δεν καλύπτονται από ε, τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία, δηλαδή τι συμβαίνει στον ψηφιακό πλανήτη. Και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να βελτιώσουμε ε, με νέες μεθοδολογίες χαρτογράφησης και θα σας δώσω κάποιο παράδειγμα για να καταλάβετε πώς το κάνουμε. για τα μουσεία που αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής μας ε, ε κληρονομιάς. Το ΕΓΜΟΥΣ είναι μια οργάνωση που δεν θα τη χαρακτηρίσω καν οργάνωση, είναι μια μικρή ομάδα ατόμων που εθελοντικά εργάζονται και συλλέγουν στοιχεία για τα ευρωπαϊκά μουσεία. Αρκετά λεπτομερή στοιχεία. Και η συλλογή αυτή είναι αρκετά εναρμονισμένη. Για παράδειγμα, στοιχεία που μπορούμε να βρούμε στην ιστοσελίδα τους είναι ο αριθμός των εθελοντών ως ποσοστό συνολικού προσωπικού, που είναι πολύ καλός δείκτης για να μπορεί κανείς να ε, υπολογίσει το μέγεθος του κλάδου πέραν όσων αμείβονται επισήμως. Επίσης, αριθμός επιδοτήσεων ως ποσοστό συνολικού εισοδήματος, επίσης καλός δείκτης για να μετρηθεί η εξάρτηση των μουσείων από τις δημόσιες ε, ε, επιδοτήσεις. Επίσης, έχουμε κάποιες πηγές που μας ε, επιτρέπουν να κάνουμε ε, κάποιους υπολογισμούς. Αυτό το γράφημα είναι από το Google που είναι οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο για παραστάσεις και παραστατικές τέκνες. Βλέπετε πως οι αναζητήσεις αυτές έχουν μειωθεί. Δεν ξέρουμε γιατί, χρειάζεται εδώ να γίνει έρευνα, αλλά το βασικό που μας ενδιαφέρει είναι πως δεν πρόκειται για στοιχεία τα οποία μπορεί να βρει κανείς τα επίσημα στατιστικά δεδομένα, αλλά είναι ένας καλός δείκτης για να μετρήσουμε το ενδιαφέρον που υπάρχει για τον πολιτισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αν δούμε ποια είναι η διείσδυση του διαδικτύου, θα δείτε πως επιταχύνεται συνέχεια και με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να μελετήσουμε τον πληθυσμό, το ποσοστό του πληθυσμού μάλλον, που ασχολείται και μπορεί αυτό το νούμερο να είναι υψηλότερο από αυτό που θα ε, μας δώσει μια πιο παραδοσιακή πηγή πληροφόρησης. Για τη βελτίωση των επισήμων ε, στατιστικών δεδομένων θα σας δώσω ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι μια νέα μεθοδολογία χαρτογράφησης και χρησιμοποιεί επίσημα δεδομένα και στοιχεία από το διαδίκτυο για να εντοπίσει επιχειρήσεις, ε, για παράδειγμα από τον κλάδο των παιχνιδιών βίντεο. Δηλαδή έχουμε 600 εταιρείε οι οποίες εντοπίστηκαν μέσω αυτής της ε, τεχνικής που είναι το web scraping που είναι σάρωση του διαδικτύου και αυτό συγκρίνεται με τα αρχικά στοιχεία που έχουμε από τα, σημαντικά, από τα ε, επίσημα ε, δεδομένα, εκεί είχαμε 1320 και το 90% αυτών των εταιριών που εντοπίσαμε μέσω ε, αυτού του web scraping είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι μπορεί έτσι να βρούμε ένα τρόπο για να εντοπίσουμε ποιες είναι αυτές οι εξαιρετικά μικρές επιχειρήσεις που δεν ε, μπορεί κανείς να βρει μέσω των επισήμων δεδομένων. Δεν αποτελεί πανάκια βέβαια αυτό τούτου είδους η συλλογή εναλλακτικών δεδομένων, καταρχήν για τη δημογραφική κάλυψη, γιατί δεν καλύπτουν ε, όλα τα 28 κράτη-μέλη. Σε γεωγραφικό επίπεδο, αν δείτε τι κάνει το ΕΓΜΟΥΣ, θα δείτε πως προσπαθούν να καλύψουν και τα 28 κράτη-μέλη, αλλά αν δείτε πιο λεπτομερώς τα στοιχεία τους, θα δείτε πως έχουν πολλά κενά από τη μια χρονιά στην επόμενη για τα διάφορα κράτη. Και βεβαίως υπάρχει το θέμα της συγκρισιμότητας και της ποιότητας των δεδομένων, γιατί δεν ακολουθούν απαραίτητο τα ίδια πρότυπα, τα οποία είναι απαραίτητα για να συλλέξει κανείς επίσημα στατιστικά στοιχεία. Παρ' όλα αυτά, δεδομένων των περιορισμών που έχουμε και με τα επίσημα δεδομένα και με τα αναλλακτικά, ο μόνος τρόπος να έχει κανείς μια καλύτερη κατανόηση, πιο σφαιρική κατανόηση του κλάδου, είναι να τα χρησιμοποιήσουμε με συμπληρωματικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη ε, τους περιορισμούς αμφωτέρων. Τώρα, στις συστάσεις μας. Ακολουθήσαμε μια σειρά από βασικές αρχές. Η συλλογή δεδομένων, όπως γνωρίζετε, είναι εξαιρετικά δαπανηρή. Προσπαθήσαμε λοιπόν να παρουσιάσουμε συστάσεις με βιώσιμες ε, δράσεις λόγω των οικονομικών περιορισμών και να βασιστούμε και σε εργασίες που έχουν γίνει και γίνονται αυτή τη στιγμή από τη Eurostat και από την σχετική ομάδα εργασίας και να κλείσουμε τα κενά κινητοποιώντας όλες τις πηγές που έχουμε διαθέσιμες και δημιουργούνται κάποιες λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν και βραχυπρόθεσμα αλλά και λίγο πιο φιλόδοξες που μπορούν να, μπουν, ε, να δρομολογηθούν μακροπρόθεσμα. Έχουμε εδώ λοιπόν τις πιο βασικές συστάσεις. Καταρχήν προτείνουμε να συλλέγονται τα δεδομένα λαμβάνοντας υπόψη τους οικονομικούς περιορισμούς και κυρίως να συλλέγονται δεδομένα για τις πολιτικές προτεραιότητες που έχουμε και δώσαμε κάποια παραδείγματα που είναι για παράδειγμα η πολιτιστική διαφορετικότητα, η πολιτιστική συμμετοχή. Επίσης να ενημερώνουμε τα στατιστικά ε, τους στατιστικούς δείκτες ταξινόμησης έτσι ώστε να είναι αντιπροσωπευτικοί στατιστικά μιλώντας του κλάδου να στοχεύσουμε στους κλάδους οι οποίοι δεν καλύπτονται αρκετά, για παράδειγμα πολιτιστικά, σχέδιο, μόδα και για αυτά να δημιουργήσουμε τη συγκεκριμένη μεθοδολογία που θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε τι γίνεται και ψηφιακά. Και τέλος, το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου να ε, χρησιμοποιήσουμε τα big data για να μπορέσουμε να σαρώσουμε το διαδίκτυο και να μαζέψουμε όγκο στοιχείων για την ψηφιακή οικονομία. Με τρεις τρόπους θα τα εφαρμόσουμε αυτά. Έχουμε το βασικό σενάριο που είναι χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα εργασίας ε, της Eurostat με επέκταση αυτού μετά το 2018 γιατί κανονικά εκεί τελειώνει και ολοκληρώνει τις προσπάθειες που κάνει. Δεύτερο σενάριο, πιο φιλόδοξο και κάπως πιο δαπανηρό. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ε, συνεργαστούν με εναλλακτικέ πηγές για να βελτιώσουν την ε, ποιότητα των δεδομένων τους με μια ενιαία πλατφόρμα έτσι ώστε να δημιουργήσουμε και ένα κοινό αφήγημα για τους πολιτικούς κλάδους στην Ευρώπη και τέλος προτείνουμε να δημιουργήσουμε και ένα διοικητικό συμβούλιο για την ε, δημιουργική ηγεσία που θα βοηθήσει στην συλλογή των δεδομένων. Να παρουσιάσω τέλος το πιο φιλόδοξο σχέδιο είναι η σύσταση ενός κατάλληλου παρατηρίου που θα συμπληρώνει τις προσπάθειες που κάνει και το παρατηρητήριο για τα οπτικοακουστικά στην Ευρώπη αλλά και η Eurostat. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Σας ευχαριστούμε. Προφανώ εγώ θα προτιμούσα την φιλοδοξότερη επιλογή σε ό,τι με αφορά. Μπορεί βεβαίως να υπάρξει και μια ενδιάμεση κατάσταση, αλλά καλό θα ήταν να ξεκινάμε φιλόδοξα. Σας ευχαριστώ πραγματικά για τις παρουσιάσεις σας και την ε, Eurostat και την ΕΑΚ ε, και τον Γενικό Διευθυντή Τζαμπιέρη για ε, αυτή την παρουσίαση. Έχουμε μια σειρά από ραντεβού που δεν πρέπει να χάσουμε την προετοιμασία του προπολογισμού 2017 κυρίως ε, εν ώψη αυτής της διαδικασίας και πρέπει όλες οι σχετικές συζητήσεις να γίνουμε για να είμαστε πιο συνεπείς με τους στόχους μας για την παιδεία και τον πολιτισμό. Έχουμε την έκθεση εκτέλεσης των προγραμμάτων. Εκεί θα πρέπει λοιπόν να επαληθεύσουμε και κάποιες νέες προσεγγίσεις και βεβαίως η βάση δεδομένων σας σίγουρα θα εμπλουτιστεί Επίσης θα φροντίσουμε να υπάρξει μια έκθεση για τη βιομηχανία της δημιουργίας και του πολιτισμού και πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα οι για τα νέα πρότυπα, τα νέα μοντέλα και την διεύρυνση του φάσματος. Απλώς εδώ γύρονται δύο ερωτήματα. Πρώτον, αυτό είπε και ο δόκτωρας Μέρση και τη συγκρισιμότητα, την αξιοπιστία και την ε, ε, τεκμηρίωση των δεδομένων και απ' την άλλη ότι πρέπει όλα αυτά να λαμβάνονται υπόψη και στους δείκτες ευημερίας, κάτι που δεν πρέπει να παραβλέπουμε. Δεν θέλω λοιπόν να στερήσω χρόνο ομιλίας από τους συναδέλφους. Έχουν ζητήσει κάποιοι το λόγο. Πρώτος ο συνάδελφος Ντρογεύσκη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας. Από το 2007 έψαχνα στατιστικά δεδομένα και πρέπει να πω ότι αυτό που βρήκα για την περίοδο 2007-2010 ήταν τουλάχιστον μη ικανοποιητικό από την άποψη της μεθοδολογίας και της πρόσβασης στα δεδομένα. Η Πολωνική Προεδρία το 2011 όταν ήμουν υπουργό ε, Πολιτισμού έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην βελτίωση της συλλογής δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλω λοιπόν να σας συγχαρώ για τα όσα πετύχατε. πολλοί μεθοδολογικοί φραγμοί έχουν πλέον αρθεί. Γνωρίζω ότι η κατάσταση δεν είναι ακόμη πλήρως ικανοποιητική Έχουμε όμως ένα πλήρες ε, σύνολο δεδομένων για το διάστημα 2010-2011, όχι όμω για το 2013-2014. Υπάρχουν ελλείψεις από συγκεκριμένε χώρες. Οι χώρες αυτές ακριβώς δεν απαντούν ε, στις ερωτήσεις όπως θα θέλατε και δεν έχετε και τρόπο να τις εξαναγκάσετε. Γνωρίζω επίσης, πέραν αυτών των περιορισμών σας, ότι υπάρχει πρόβλημα με την κατηγοριοποίηση των ε, δαπανών. Στην Γερμανία, λόγω χάρη, ένα πρόγραμμα μαγειρική στην τηλεόραση, μια εκπομπή μαγειρική στην τηλεόραση, θεωρείται πολιτισμό. σω γιατί είναι άχρηστη στη μαγειρική η Γερμανία. Στη Γαλλία ή την Ιταλία όμω τα προγράμματα μαγειρική θεωρούνται εμπορικέ εκπομπέ. Το γεγονός είναι ότι στις στατιστικές, στατιστικά δεδομένα του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα στυλό και τα μολύβια θεωρούνται δαπάνη για τον πολιτισμό, ενώ σε κάποια κράτη όχι. Παρόμοια προβλήματα υπάρχουν με τα video games στους υπολογιστές και το σχετικό του εξοπλισμό. Δεν θα ήθελα όμως να χάσω την ευκαιρία να σας συγχαρώ για τα όσα πετύχατε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό που με ενδιαφέρει όλος ιδιαίτερος είναι να καλυφθούν τα κενά. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες σας αυτή τη στιγμή για το 2016. Και τι αναμένετε από τις εκθέσεις που έρχονται ένα πενταετία στα χέρια σας. Ποια είναι τα κάτι μελη που περισσότερο καθυστερούν ή δεν συνεργάζονται στην υποβολή δεδομένων όπως τα ζητάτε. Επίσης κυρία Κώστα να πω ότι πολύ θα ήθελε να συντάξω μια έκθεση για το κόστος της πολιτιστικής συμμετοχής και με ενδιαφέρει πολύ ποιε χώρες έχουν το, καταβάλουν το υψηλότερο κόστος για τη συμμετοχή σε πολιτιστικέ δραστηριότητε, ιδίω τους, για τους πολίτες με χαμηλά εισοδήματα. Ευχαριστώ συνάδελφε. Εξαιρετική ανάλυση αυτή που κάνατε στην παρουσίασή σα, ο κύριος Μόργανο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση από καρδιάς ε, και ευχαριστούμε την Eurostat γιατί πραγματικά αυτά τα βήματα πρόοδου μας επιτρέπουν να προωθήσουμε και τις πολιτικές μας αναζητήσεις. Οι απαιτήσει αφήνειας για τον όρο πολιτισμό και ό,τι αυτό συμπεριλαμβάνει ήταν ε, πολύ εύστοχες. Επίσης η έκκληση για το ποσοστό προς το, το σύνολο της απασχόλησης και αυτό είναι σημαντικό γιατί το 29,2% ε, είναι ένα μεγάλο ποσοστό ακόμη και σε σχέση με τις δραστηριότητες της Επιτροπής μας και μια μελέτη που θα χρειαστεί να γίνει προς την κατεύθυνση περισσότερης απασχόλησης αλλά περισσότερης απασχόλησης που αξιοποιεί καλύτερα και με τρόπο ε, όσο δυνατόν πιο ε, συνολικό και τον τομέα της ψυχαγωγίας και του πολιτισμού με την αξιοποίηση όλων μας των πτυχιούχων. Επίσης, ε, η οικονομική διάσταση. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά, διότι όταν θα συζητήσουμε θέματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, ε, πολλοί πιστεύουν ότι, πρόκειται για μια, ότι συζητάμε για δαπάνες που είναι κάπως περιτές ή δαπάνες πολυτελείας. Όμως ε, ισχύει το αντίθετο και αυτό που δείχτηκε νομίζω σήμερα το πρωί, ότι πρέπει να υπάρξουν σοβαρότερες αποφάσεις για μια γραμμή που μου φαίνεται πραγματικά ότι τη συμμεριζόμαστε όχι ε, μόνο εμείς της Επιτροπής Πολιτισμού. Τώρα, για την συγκέντρωση δεδομένων σε διεθνές επίπεδο θα μας επέτρεπε αυτό να δώσουμε προσοχή και στις διάφορες ε, αντιλήψεις που υπάρχουν ανά τον κόσμο και ξέρουμε τι απαιτήσει μπορεί να υπάρχουν ε, μετά από συμφωνίες που έχουν συναυθεί σε διεθνές επίπεδο και την κυκλοφορία δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, γιατί πήρα το λόγο. Η διαδικασία που έχει ξεκινήσει να συνεχίσει και με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στις διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες, στις προσφορές του πολιτισμού. Επίσης πρέπει να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια για να βγούμε από το λεγόμενο παραδοσιακό τρόπο Εδώ χρησιμοποίησατε πραγματικά με νέα διάσταση το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το διαδίκτυο αλλά και το πόσα στοιχεία μας διαφεύγουν. Και εάν κοιτάξουμε τα πράγματα προσεκτικά βλέπουμε ότι οι νέες γενιές ταξιδεύουν περισσότερο έτσι. Όμως ο στόχος είναι να βοηθήσουμε περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη διάσταση του πολιτισμού και των ε, σχετικών βιομηχανικών, βιομηχανιών και κλάδων. Πρέπει να δούμε πού στοχεύουν οι παρεμβάσεις μας και να εξισορροπήσουμε καλύτερα τα πολιετή δημοσιονομικά προγράμματα. Λόγω χάρη αυτό ο αριθμό των 600 επιχειρήσεων που το εντοπίσατε μέσα από αυτή την μέθοδο μου φαίνεται ένα πολύ σημαντικό στοιχείο κατάλαβα ότι γίνεται προσπάθεια για περαιτέρω διευκρίνηση της μεθοδολογίας σας. Όμως, για τα θέματα αυτά που αντικειμενικά είναι καινούρια και είναι πρωτοποριακά, δεν πρέπει να φοβόμαστε. Πρέπει να βγαίνουμε από τους ε, κανόνες και από την πεπατημένη, αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε Λουίντι Η κυρία Γκριμπάτσκα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι ευγνώμων για αυτήν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Το μέλλον, στο μέλλον θα είναι πολύ καλό να έχουμε βρει την απάντηση στην ερώτηση, στο ερώτημα σε πιο εύρος η χρήση του διαδικτύου οδηγεί σε μείωση όσον αφορά την κατανάλωση του υλικού πολιτισμού. Ελπίζω λοιπόν ότι όσα και να μπορεί να βρει κανείς στο διαδίκτυο θα υπάρχουν, θα υπάρχουν πάντα οι πολίτες που θα ενδιαφέρονται να επισκεφθούν μουσεία για να δουν τις συλλογές τους και να τις απολαύσουν. Νομίζω ότι μπορεί να ανοιχνεύσει κανείς σαφείς τάσεις από τα στοιχεία αυτά και δεν θα πρέπει να φοβηθεί κανείς ε, να συναγάγει κάποια συμπεράσματα. Είναι λοιπόν ζωτική σημασίας στην παιδεία και εκπαίδευση των πολιτών να καλλιεργήσουμε την κατανάλωση πολιτιστικών και πολιτισμικών προϊόντων Διαφορετικά θα καταλήξουμε σε πολίτες οι οποίοι θα συλλέγουν κάποια πληροφοριακά στοιχεία αλλά δεν θα συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις πολίτης. Ευχαριστούμε για την κέρια παρέμβασή σου Κριστίνα. Ε, δεν υπάρχουν άλλοι συναδελφοί. Να πω λοιπόν ότι εδώ μόλις ανοίξαμε ένα διάλογο για τα θέματα αυτά. Θα σας ξαναδώσω το λόγο για να απαντήσετε και αν θέλετε να συμπληρώσετε κάποιες παρατηρήσεις που δεν προλάβατε προηγουμένως. Πάντως όπως ε, μιλήσαμε και για την Δημιουργική Ευρώπη. Είναι σημαντική η μελέτη αντικτύπου που ετοιμάζεται για να μπορούμε ε, έπειτα να αποφασίσουμε από κοινού πώς ε, θα δώσουμε συνέχεια σε όλα αυτά και βάσει των ενδείξεων που προέκυψαν τι κατεύθυνση θα δώσουμε για να δούμε τις διάφορες επιλογές και να δούμε πώς θα κινηθούμε. Να σας δώσω το λόγο με τη σειρά που εσείς νομίζετε. Ίσως ανάποδα να πάρετε το λόγο. Se vuole aggiungere Valentina Montaldo e Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ για τις ευχαριστίες σας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ήταν τόσες πολλές οι τεχνικού χαρακτήρα ερωτήσεις. Ένα ή δύο στοιχεία από πλευράς μου η συμμετοχή των κρατών μελών στη συλλογή αυτών των δεδομένων δεν είναι μια εναλλακτική εθελούσιου, εθελοντικού χαρακτήρα δραστηριότητα, είναι υποχρεωτική δραστηριότητα αυτή η συμμετοχή. Υπάρχουν κανόνες και κανονισμοί που αφορούν τα κράτη-μέλη και δεσμεύονται να μεταδίδουν, να δίνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά τα στοιχεία υποχρεωτικού χαρακτήρα συλλογή ε, στοιχείων που πρέπει να συλλέγονται υποχρεωτικά από τα κράτη-μέλη. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την ποιότητα και αξιοπιστία αυτών των στοιχείων σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Εξ άντε, εκ εργαζόμαστε ώστε να μπορούν να ε, αντιμετωπίζουν και να καλύπτουν ε, τα, τις ανάγκες ε, ε, συλλογής στοιχείων, συγκρίσιμων στοιχείων μεταξύ τους. Κάνουμε λοιπόν εκ προημίου έργο ώστε να συλλέγονται με συγκρίσιμο τρόπο αυτά τα στοιχεία, να είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους. Αυτό σε σχέση και με την αποσαφήνιση για τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται η Eurostat, η Eurostat όσον αφορά την συμμετοχή στα πολιτιστικά και πολιτισμικά και το διαδίκτυο και την αποϊλοποίηση ως ε, διάσταση δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την πραγματικότητα του διαδικτύου ως ενός στοιχείου για την διάδοση όχι μόνο για την αγορά αγαθών αλλά και την διάχυση δεδομένων και στοιχείων. Και εδώ υπάρχει δυνατότητα να γίνουν περισσότερα, να γίνονται περισσότερα ως προς αυτή τη διάσταση. Για να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την τόσο θετική αντίδραση που είχατε και δύο σημεία στα οποία θα ήθελα να σταθώ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό καταρχήν για τις ε, συστάσεις τις ίδιες. Νομίζω ότι οι προτεραιότητες για τη συλλογή δεδομένων αποτελούν ένα θέμα γιατί πολλές φορές αλλάζουν και οι πολιτικές προτεραιότητες και οι μηχανισμοί οι οποίοι είναι ε, οικονομικοί για τη συλλογή δεδομένων δεν είναι τόσο εύκολο να δημιουργηθούν. Και τόσο από ο κύριος Μόργανο οι εναλλακτικέ ε, πηγέ δεδομένου ποτέ δεν θα έχουν την ίδια ποιότητα και συγκρισιμότητα με τα δεδομένα τη Eurostat. Αλλά δεν θα πρέπει όμω να φοβόμαστε και νέε μεθοδολογίε για τη χρήση των ε, big data που γίνεται online. Γιατί ο ίδιος ο κλάδος αυτή τη στιγμή εξελίσσεται με νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες αλλά και με νέους τρόπους συμμετοχής ε, στον πολιτισμό. Οπότε είναι και αυτό ένα στοιχείο. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω και σας ευχαριστώ για το ότι με ακούσατε. Είναι όντως για μας μια προτεραιότητα. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που για σας ισχύει αυτό. Τα στοιχεία τα οποία έχετε δει μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χάραξη πολιτικής. Αυτά τα δεδομένα χρειαζόμαστε έτσι και αλλιώς. Και όταν λέμε πως ο πολιτισμός βρίσκεται στην ε, καρδιά της οικονομίας της γνώσης, έχουμε πια τα στοιχεία που το τεκμηριώνουν για όλα τα ε, κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν λέμε ότι θα πρέπει στην ψηφιακή ενιαία αγορά να βρίσκεται στην πυρήνα αυτής ε, ο πολιτιστικός κλάδος, νομίζω ότι και αυτό πλέον αποδεικνύεται. Στοιχείο πολύ σημαντικό για τη συμμετοχή στα πολιτιστικά. Έχουμε στοιχεία τα οποία όλα γνωρίζαμε τα οποία όμως δεν ξέραμε ε, τι μέγεθος έχει το πολιτικό χάσμα για θέμα κοινωνικής συνοχής, για θέμα οικονομικό, για το γεγονός πως πάρα πολλοί μένουν πίσω. Για το διαδίκτυο. Οι συνάδελφοι εξήγησαν πόσο δύσκολο είναι να έχει κανείς συγκεκριμένα στοιχεία για την εμπορία υπηρεσιών. Γιατί αυτή τη στιγμή Έχουμε το streaming, έχουμε τα ηλεκτρονικά βιβλία, τα e-book. Οπότε αυτή τη διάσταση σε διεθνέ επίπεδο πολύ δύσκολο να την παρακολουθήσει κανεί. Έχουμε κάποια στοιχεία περιστασιακά, δηλαδή ε, κάποια πουλιούνται, ε, ας πούμε, ε, e-book, λιγότερα από τα βιβλία σε χαρτί. Εντάξει, αυτό μπορεί κανείς να το πει τώρα για τα μουσεία τα οποία έχουν ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρουν στο κοινό τους. Ε, το περίεργο είναι ότι παρόλο που υπάρχει αυτή η ψηφιακή δυνατότητα επίσκεψης δεν έχει μειωθεί η συνολική επισκεψιμότητα στα μουσεία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει τρόπο συνδυασμού ε, των δύο ε, τύπων επισκεψιμότητας. Γιατί τα εναλλακτικά στοιχεία, δεδο... τις εναλλακτικές πηγές δεδομένων τα παρακολουθούμε και διαπιστώνουμε ότι αυτό που σας είπα για τα μουσεία ισχύει. Για την πολιτική, τι μπορούμε να κάνουμε με τα υπόλοιπα ε, δεδομένα που προκύπτουν από εναλλακτικέ πηγές. Καταρχήν, όντω είναι εναλλακτικέ. Γιατί το, η βασικός μας, ε, το βασικό μας μέλημα θα πρέπει να παραμείνει η συλλογή μέσω Eurostat από όλα τα 28 κράτη-μέλη. Επίσης υπάρχει μια διαδικασία που βοηθά τα κράτη-μέλη να βελτιώνουν ε, και τα δικά τους δεδομένα. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δηλαδή. Ακόμα ε, έχουν υποεκτιμηθεί κάποια από τα στοιχεία γιατί δεν συλλέγουν όλα τα κράτη-μέλη με την ίδια ακρίβεια τα σχετικά στοιχεία. Και το λέω αυτό και ως ε, εμπειρογνώμονας αλλά και ως άνθρωπος ο οποίος τα καταναλώνει τα στοιχεία αυτά. Για το παρατηρητήριο, ίσως είναι υπερφιλόδοξο δεδομένου του πλαισίου στο οποίο κινούμαστε το να δημιουργεί ένα παρατηρητήριο, είναι εξαιρετικά δαπανηρό και τα χρήματα θα πρέπει να προέρχονται από το ε, Creative Europe, το οποίο μοιάζει μεγάλο πρόγραμμα, αλλά δεν είναι. Έχει πολλαπλές λειτουργίες και ο πιο βασικός στόχος είναι η συνεργασία μεταξύ project, τα δίκτυα, η συνεργασία διασυνοριακή σε πολιτιστικό επίπεδο. Οπότε είναι μια συζήτηση την οποία θα πρέπει να συνεχίσουμε ε, στο μέλλον. Για το δεύτερο εναλλακτικό σενάριο εκεί υπάρχουν πολλά στοιχεία που μας ενδιαφέρουν. Και βεβαίως ε, με χαρά συναντάμε και τον κλάδο και παίρνουμε τα στοιχεία που έχει, αλλά υπάρχει μια σύσταση η οποία δεν μας ικανοποιεί. Το δηλαδή θα πρέπει να ξεκινήσουμε με τους κλάδους στους οποίους έχουμε πολύ λίγη πληροφόρηση. Δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι παραγωγικό. Είναι ως ιδέα πολύ θετικό σε ένα ιδανικό κόσμο ξεκινάς από εκεί που έχει δυναμίε και χτίζει πάνω σε αυτό. Αυτό το οποίο σκεφτόμαστε, γιατί πιστεύω ότι αυτό που προτείνεται δεν θα λειτουργήσει, είναι να ξεκινήσουμε με τους κλάδους στου οποίου στους οποίους είναι η καλύτερη κατάσταση, δηλαδή μουσική. Γιατί εκεί στον κλάδο αυτό υπάρχουν δεδομένα και είναι πιο εύκολο να κάνουμε πρόοδο και να αποδείξουμε ότι αυτό που κάνουμε έχει σημασία. Γιατί αν ξεκινήσουμε με ένα πολύ αδύναμο κλάδο, μετά από τρία χρόνια θα έχουμε καλύψει ένα πολύ μικρό ποσοστό και αυτοί οι οποίοι θα αποφασίσουν τον προπολογισμό για το επόμενο πρόγραμμα θα μα πούνε γιατί να συνεχίσετε. Άρα λοιπόν θα ξεκινούσαμε μάλλον με ένα κλάδο ως αυτός της μουσικής που υπάρχει στα στοιχεία μας και βεβαίως το θέμα αυτό θα το ξανασυζητήσουμε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ίσως και μέσω κάποιου ε, πειραματικού έργου, ένα pilot project δηλαδή, αν και εσείς το επιθυμείτε. Thank you. Ευχαριστώ. Είναι πολύ ε, ενδιαφέρουσα πιθανότητα προκειμένου να μην δοθεί το μήνυμα ότι με, βάζουμε όλους τους κλάδους στο ίδιο επίπεδο. Ότι δεν βάζουμε μάλλον του κλάδου, κύριε Πρόεδρε. Κύριε το λόγο. Θα ήθελα να. Η Χέλγα, θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα αυτό για τι επεξηγήσει. Σα είπατε ότι σα ικανοποιεί ότι υπάρχουν στοιχεία να δείξουν την τεράστια επίπτωση αυτής της βιομηχανίας στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η επίπτωση όλων αυτών που γνωρίζουμε και που μπορούμε να δείξουμε σε σχέση με την Επιτροπή και την προσέγγιση για την ενιαία εσωτερική αγορά που αφορά σε κάποιο βαθμό και τις εξωτερικές μας σχέσεις και την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Βλέπετε ήδη λοιπόν κάποιες μεταθέσεις ε, όσον αφορά τις προσδοκίες, το τι αναμένεται να ακολουθήσει τώρα. Ευχαριστώ. <laughs> Well, I don't want to be over... Να απαντήσετε αν μπορείτε. Δεν θέλω να είμαι υπεραισιόδοξος. Η κατεύθυνση όμως σε σχέση με αυτή την αγορά δεν θα πρέπει να αποτελεί κάποια ανησυχία για τον τομέα του πολιτισμού. Συμμετείχαμε σε στις δραστηριότητες αυτές ευθύς εξ αρχής πάντα και νομίζω τα αποτελέσματα είναι αρκετά καλά συνολικά σε όλο αυτό το εύρος δραστηριοτήτων και στην προσοχή που στρέφουμε στο διαδίκτυο και σε σχέση με τις τάσεις αυτές και αν θέλει κανείς να αποδείξει τις επιπτώσεις αυτές έχουμε τις επιπτώσεις τα κέρδη που συνεπάγεται αυτή, συνεπάγονται οι δραστηριότητες αυτές θα ήθελα λοιπόν να πω σε σχέση με τις, ε, ε, ε, την αναθεώρηση όσον αφορά. Αυτή δεν λέει πάρα πολλά για τον πολιτισμό. Θα έπρεπε να έχουμε τα στοιχεία και χρησιμοποιούμε το διμερές πλαίσιο για μια πολιτιστική πολιτική με τους εταίρους μας. Η Τινησία είναι το πρώτο παράδειγμα. Τα πράγματα βαίνουν αρκετά καλά και σε σχέση με την Creative Europe και τις χώρες που συμμετέχουν δημιουργούμε αυτό το πλαίσιο που βοηθούμε να αναπτυχθούν οι δυνατότητες και το δυναμικό των χωρών εταίρων και τους παρέχουμε τις ευκαιρίες να συμμετάσχουν μέσα στις πολιτισμικές αυτές δραστηριότητες της Ευρώπης. Από κοινού κάνουμε αυτό το, ε, αυτή την, το έργο ακολουθούμε με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πράγματα βαίνουν αρκετά καλά μπορώ να πω. Και μια ερώτηση που έγινε για το εμπόριο. Δεν είναι τόσο πολύ οι συμφωνίες εμπορίου για το τι επιθυμεί κανείς να κάνει. Έχουμε μια θέση για το εμπόριο με τις ε, ανταλλαγές και τις ε, επαφές ε, όσον αφορά τον πολιτισμικό τομέα μπορούμε να προχωρήσουμε πιο πέρα. Δεν κάνουμε λόγο για κάποιες ευρύτερες αλλαγές. Είναι ένα θέμα το οποίο συμμετέχει, εντάσσεται σε αυτές τις εξελίξεις για το τι θα μπορούσε να γίνει μελλοντικά όσον αφορά τον πολιτισμικό τομέα. Το είπε η κυρία Κώστα στην αρχή. Θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό και το έργο όσον αφορά την ε, Βαλεντίνα δεν έγινε με απομονώ σε κάποιο στεγανό. Συμμετείχαμε ευθύ εξ αρχής ε, και οι γενικές μας διευθύνσεις ε, με την εμπλοκή τους παρακολουθούν αυτά τα πράγματα. Είναι λοιπόν κάτι που παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι συμμετέχουμε σε αυτό το πλαίσιο και είμαστε αισιόδοξοι. Το ελπίζουμε και εμείς διότι εδώ νομίζω όλοι πραγματικά έχουμε περίπου τις ίδιες ανησυχίες. Στην αρχή η αίσθηση που είχαμε είναι ότι τα επιχειρήματα που προβάλλονταν και τα αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιούνταν για το τι σημαίνει εισαγωγή και εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών αλλά κυρίως για τους δείκτες της ανώτατης εκπαίδευσης, της πολιτιστικής συμμετοχής Ο δεσμός, η σχέση μεταξύ της απασχόλησης και του πολιτισμού, η βελτίωση της πορείας και του ΑΕΠ, όλα αυτά δείχνουν πράγματα που δεν σημαίνει ότι από την Επιτροπή αξιολογούνται όπως θα έπρεπε. Αυτή νομίζω ήταν κάπως ε, η ερώτηση που έκανε η κυρία Τρούπελ. Άλλωστε, μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στην στρατηγική για την ενιαία ψηφιακή αγορά στο δεύτερο μέρος της συζήτησης, διότι στην αρχή η έμφαση στην πνευματική ιδιοκτησία και στα πλαίσια της ενιαίας ψηφιακής αγοράς είναι εάν όχι ανεπαρκής αλλά νομίζω το Κοινοβούλιο και η Πολιτιστική Επιτροπή επεδίωξε διαφορετικά αποτελέσματα. Θέλουμε να υπάρξει φιλόδοξη στρατηγική πολιτιστικής δημοκρατίας όπως ανακοινώθηκε και νομίζω ότι εδώ έχουν επιμείνει τουλάχιστον τρεις ε, επιτροποί πέραν της Πρόεδρου της Επιτροπής Στοιχείο βασικό λοιπόν εδώ είναι να συνδέσουμε την λέξη growth, οικονομική ανάπτυξη, με τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Δεν είναι ε, αυτονόητο. Όμως για να υπάρχουν θέσεις απασχόλησης ποιότητας, ε, η εκπαίδευση που να σχετίζεται και με την πολιτιστική αξία και η κοινωνική ένταξη αλλά και η ανάπτυξη μέσω του πολιτισμού είναι στοιχεία που χρήζουν διεπιστημονικής προσοχής από την Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε πάντως ε, όλους γιατί η δουλειά σας ήταν, ε, είναι κέρια και πιστεύουμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να δώσουμε φωνή και να αποδείξουμε ότι η πολιτιστική διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών ε, είναι πολλά υποσχόμενη. Είναι και κυκλική, διότι αποδείχθηκε ότι σε καιρούς κρίσης, όταν πέφτουν όλοι οι δείκτες, προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία περί ανθεκτικότητας Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό για την πολιτιστική διάσταση. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από αυτή τη συνάντηση και έγραφα θα υπάρξουν ε, για όποιον ενδιαφέρεται εφόσον υπάρχει αυτή η κοινή διάθεση να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ την Eurostat για όλη τη δουλειά και θα θέλαμε να καταλάβουμε και από την άποψη των πόρων εάν σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι συνεπής προς την επένδυση αυτή και να αφήσει χώρο και για πρόοδο, γιατί χωρίς τέτοιες ενδείξεις είναι δύσκολο να καταλάβουμε πού ε, οδεύει ο πολιτισμός και η πολιτιστική παραγωγή. Πραγματικά λοιπόν ευχαριστούμε, κλείνουμε αυτό το πάνελ και ξέρουμε ότι έχει ήδη φτάσει ο επόμενος ε, συζητής μας, ο επόμενος προσκεκλημένος. Οπότε δύο λεπτά ε, διάλειμμα για να χαιρετηθούμε και μετά θα συνεχίσουμε. Sorry, please, we, we continue our... Συνεχίζουμε λοιπόν συνάδελφοι. Uh, silence please. Λίγη ησυχία παρακαλώ. Excuse me, can you take your seat please? Καθίστε παρακαλώ, ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τις εργασίες μας. And so? Allora, eh, ora abbiamo una interessante ε, ε, eh, έχουμε μια ενδιαφέρουσα ακρόαση με τον Στέφανο Ντομινιόνι τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για τους Πολιτιστικούς Δρόμους του Συμβουλίου της Ευρώπης. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, περιμένουμε να έχουμε την προσοχή σας. Ξεκινήστε παρακαλώ. Ωραία. Ε, Έλεγα ότι θα ξεκινήσουμε να ακούσουμε τον κύριο Ντομινιώνη που είναι διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τους πολιτιστικούς δρόμους του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Λουξεμβούργο και όπως τα ξέρετε αύριο τα διαπολιτιστικά προγράμματα κλείνουν 30 χρόνια. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ακόμα από τώρα του τους ερωτισμούς μας. Έχουμε 33 διαδρομές ε, πολιτιστικές στην Ευρώπη στην Ευρώπη ξεκίνησαν αυτά τα προγράμματα και υπάρχουν σημαντικέ μορφέ συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων με εταιρικέ σχέσεις ή με μερικές ή διευρυμένε διμερείς συμφωνίες. Επίσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέρετε ότι οι πολιτιστικέ διαδρομές συμπεριλήθησαν και στην Δημιουργική Ευρώπη ω μία από τι ε, ενδιαφέρουσες πολιτιστικέ πολιτικές και σε αυτή τη φάση η αμοιβαία αναγνώριση, ο διαπολιτιστικός διάλογος ξεπερνούν τα σύνορα. Σύνορα που αυτή τη στιγμή κάπως ε, ούτως ή άλλως αφισβητούνται στην Ευρώπη που κλείνει τα σύνορα. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε όλες τις πολιτιστικές ε, πολιτικές που μας δίνουν μια αίσθηση του ανήκειν και μια αίσθηση ταυτότητας. Ξέρετε ότι το Ινστιτούτο του Λουξεμβούργου έχει σημαντικές ευθύνες στην υλοποίηση του προγράμματος των διαδρομών αλλά είναι και υπεύθυνο για την αξιολόγηση των προγραμμάτων και για την ε, έγκρισή τους και για να αποτιμήσει τη δυνατότητά τους να είναι πραγματικοί φορείς ε, παιδείας αξιοποίησης και να ε, υπάρξει πρόσβαση σε αυτά. Δεν διατηρούνται διαβίου αυτές οι διαδρομές, επενδύονται, βελτιώνονται και επανεκτιμώνται. Θα έχουμε λοιπόν τη χαρά να σας ακούσουμε. Σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ και θα σας δώσω το λόγο για 15 περίπου λεπτά. Και μετά θα έχουμε ερωταπαντήσεις από τους συναδέλφους. Το Παρακαλώ, δόκτωρα Δομινιώνη. Ε, ε, Κυρία Κώστα, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Είναι μεγάλη μου χαρά για το Συμβούλιο της Ευρώπης να βρίσκομαι εκ μέρους του Συμβουλίου της Ευρώπης να βρίσκομαι εδώ. Είστε φίλοι μας εδώ και χρόνια είναι φίλος επί πολλά χρόνια του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε σχέση με τα όσα έκανε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για την πρόσκλησή σας για την, να είμαστε παρόντες στην Πολιτισμική Επιτροπή είναι μια ναυαρχίδα των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, το θέμα των πολιτιστικών διαδρομών. Κατά τη δεκαετία του 80 ξεκίνησε. Είναι ένα πρόγραμμα η, τα μονοπάτια και οι πολιτισμικές διαδρομές που εξελίχθηκε επί πολλά χρόνια και έχουμε πολλές γνώσεις ε, που αποκτήσαμε από τότε μέχρι σήμερα. Με μεγάλη χαρά θα σας το παρουσιάσω λοιπόν σήμερα. οι πολιτισμικές διαδρομές. Είναι πολυεθνικά δίκτυα, διασυνοριακά δίκτυα συνδέσεων και διαδρομών όσον αφορά την, το εγχείρημα της ε, πολιτισμικής παράδοσης της Ευρώπης που συνδέει πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι εθνικού χαρακτήρα, είναι πολυεθνικού, πολυδιάστατου χαρακτήρα, πανευρωπαϊκού χαρακτήρα που συνδέει τις χώρες ε, το εγχείρημα αυτό των διαδρομών όσον αφορά τις ε, την πολιτισμική τους κληρονομιά, την ιστορία, την αρχιτεκτονική, τα, ε, την, τις τέχνες, Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε λοιπόν έτσι μια εικόνα που να σας δίνει ε, την ε, απήχηση του τοπίου, του περιβάλλοντος, των τεχνών της ίδιας της θρησκείας και πολιτισμικής παράδοσης και θρησκευτικής παράδοσης. Είναι αυτές οι ανάγκες που κάνουν τους ανθρώπους να συνέρχονται και να ε, σειραίουν σε αυτές τις διαδρομές. Είναι ένα πολυεθνικό ε, εγχείρημα που κάνει λόγο για την κοινή μας ιστορία και την κοινή μας ε, πολιτισμική κληρονομιά και παράδοση. Το Συμβούλιο της Ευρώπης λοιπόν βρίσκεται στην καρδιά, στον πυρήνα αυτού του προγράμματος. Καθορίζει τις πολιτικές και τις αξίες ε, όσον αφορά τις, ε, το, την πρωτοβουλία αυτών των διαδρομών και εντάσσονται στο καθεστώς του καταστατικού μας αυτές οι αρχές και αξίες και έχουμε την εντολή να εξυπηρετείται η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η συνεργασία στα θέματα πολιτισμού βρίσκονται ας το πω έτσι στο γενετικό αποτύπωμα αυτών των δραστηριοτήτων. Αποφάσισε το Συμβούλιο της Ευρώπης λοιπόν να δημιουργήσει ένα πυρήνα χωρών που ενδιαφέρονται σε αυτά τα, για αυτά τα προγράμματα και αυτές τις διαδρομές και μονοπάτια ώστε να προχωρήσουμε. Υπάρχει λοιπόν η συμφωνία αυτή που είναι ανοιχτή σε όλα τα κράτη και κάθε χρόνο υπάρχουν και περισσότερα που εντάσσονται και συμμετέχουν συμμετέχουν. Καθορίζεται έτσι το στρατηγικό πρόγραμμα στρατηγική σημασία για τις δράσεις αυτές και με πιστοποίηση που ε, την χάνεται και είναι μία από τις ναυαρχίδες αυτό το πρόγραμμά μας διαδρομές δηλαδή που ως παραδείγματα πιστοποιούνται και αξιολογούνται ε, σε τακτά διαστήματα και όλα αυτά βρίσκονται ε, στον ιστό αυτών των ε, δράσεων μας. Έχουμε και το θέμα και των νομικών στοιχείων που ε, αποτελούν την ραχοκοκαλιά αυτών των ε, πρωτοβουλειών ε, δράσεις νομοθετών. Θέλω εδώ να αναφέρω τρεις βασικές συμβάσεις που βρίσκονται στην απαρχή και υποστήριξη αυτών των δράσεων είναι η ε, πολιτισμική ε, σύμβαση, η παλαιότερη ε, σύμβαση όσον αφορά τις πολιτισμικές δραστηριότητες από την δεκαετία του 1950, η σύμβαση για το περιβάλλον και για την κοινωνία. Αυτές οι τρεις συμβάσεις έχουν πολύ μεγάλη εμβέλεια, διότι καθορίζουν το πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων. Συνεργασία, αλλά και συνεργασία που θα υποστηρίζει και θα εξυπηρετεί την κληρονομιά, την ευρωπαϊκή κληρονομιά με βάση τις αρχές και αξίες και εξυπηρετώντας την κοινωνία πάντα. Πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά των δραστηριοτήτων μας η εξυπηρέτηση των πολιτών και της κοινωνίας. Θα το επεξηγήσω αυτό ευρύτερα. Πρέπει στους πολίτες ακριβώς να απευθυνόμαστε ε, και έτσι δεν είναι ένα απλό ε, πρόγραμμα και πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά κάθε ομάδα διαχειρίζεται το δικό της δίκτυο και είναι υπεύθυνη για αυτό. Για να επεξηγήσω μεθοδολογικά την προσέγγιση μας αυτή πολύ σύντομα, εντάχει να σας δώσω ένα διάγραμμα του Ιδρύματος στο Λουξεμβούργο που έχουμε την έδρα μας το Γραφείο Πολιτισμικών Διαδρομών είναι η υπηρεσία που και χάρη στην υποστήριξη του Λουξεμβούργου λειτουργεί εκεί αξιολογούνται και αποτιμούνται οι διαδρομές αυτές υπάρχει συμβουλευτική δραστηριότητα για την κατάρτιση και εκπαίδευση και φυσικά και για την αξιολόγηση. Ετήσια μια ολόκληρη ένα σύνολο διαδρομών αξιολογούνται και περνούν οι συστάσει στο Συμβουλίο της Ευρώπης όπου πρέπει να επικυρωθούν, συμπληρωθούν ή ε, ε, προσαρμοστούν σε σχέση με τις ε, αρχές και τα κριτήριά μας. Υπάρχει ένας ολόκληρος κύκλος πιστοποίησης που ακολουθείται ως, ένα ας το πω έτσι πρότυπο τυποποίησης και έχουμε εδώ και τις δραστηριότητες δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης με τα βραβεία και τα διάφορα ε, έπαθλα τα οποία απονέμονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Υπάρχει και το καθεστώς υποψήφιου, υποψήφιου διαδρομής υποψήφιας να πιστοποιηθεί σε αυτό το πλαίσιο διαδρομών και ε, πολιτισμικών ε, δραστηριοτήτων και ο φάκελο, στο χαρτοφυλάκιο ε, από πλευράς υποψηφιότητας αξιολογείται από τους επαΐοντες και υποβάλλονται συστάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για το αν ή όχι μια συγκεκριμένη διαδρομή μπορεί να τύχει πιστοποίησης και να εγκριθεί και να ενταχθεί σε, ε, στις πολιτισμικές διαδρομές της Ευρώπης. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά κριτηρίων και απαιτήσεων που πρέπει σε αυτές να ανταποκρίνονται οι υποψηφιότητες για να πιστοποιηθούν Υπάρχει ένας κατάλογος αντικειμενικών κριτηρίων. Κάποια από αυτά τα βλέπετε στο γράφημα στην οθόνη σας. Οι ευρωπαϊκές αξίες έχουν τεράστια σημασία. Πρέπει λοιπόν να επικεντρώνονται αυτές οι δραστηριότητες ε, ε, σε αυτό το στοιχείο, στην κοινή πολιτισμική κληρονομιά, καλλιτεχνική κληρονομιά, ευρωπαϊκή κληρονομιά ευρύτερα. Τα κριτήρια αυτά λοιπόν συνδέονται με την έρευνα και την ανάπτυξη Πρέπει να υπάρχει λοιπόν συνεργασία που θα διασφαλίζεται στην έρευνα και ανάπτυξη για ένα συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει η Επιστημονική Επιτροπή όσον αφορά τις ε, πολιτιστικές αυτές διαδρομές που ε, εξετάζει τις ε, δραστηριότητες κατά τη διάρκεια αυτών των διαδρομών. Όμως πρέπει να υπάρχει και η εκπαιδευτική διάσταση σε αυτές τις δραστηριότητες και διαδρομές όσον αφορά τους νέους, την σχολική εκπαίδευση. Πρέπει να υπάρχει και μια ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών. Να διοργανώνονται έτσι σε τακτή βάση δραστηριότητες μέσα σε ένα πλαίσιο προγραμμάτων ώστε να μπορούν έτσι να ευθυγραμμίζονται ε, και να ε, προσαρμόζονται στις αρχές και αξίες μας αυτές οι ε, δραστηριότητες. Και ο πολιτισμικός τουρισμός είναι επίσης μια άλλη διάσταση και η αηφορία, η βιώσιμη ανάπτυξη. Βλέπουμε εδώ λοιπόν την καλλιτεχνική πολιτισμική πολιτισμική αλλά και οικονομική διάσταση που εντάσσονται, συνεντάσσονται και συνεμπλέκονται σε αυτές τις δραστηριότητες και για τις επιπτώσεις όσον αφορά το τοπικό ε, περιβάλλον να εντάσσονται και να αποβαίνουν προς όφελος και της ε, ε, οικονομίας. Πρέπει να εντάσσονται λοιπόν έτσι με αυτόν τον τρόπο ώστε να υπάρχει η βέλτιστη απόδοση. Σημαντικό είναι επίσης και το θέμα του νομικού καθεστώτος που πρέπει να συνδέεται αυτό το καθεστώς σε σχέση με μια ένωση ή σύλλογο ή μια σύμπραξη ε, τοπικών ε, δήμων, κοινοτήτων, άλλων φορέων που συνηφαίνονται σε αυτές τις δραστηριότητες. Και αυτή είναι μία από τις ε, διαφορές όχι μόνη αλλά για την πιστοποίηση αυτών των διαδρομών Πρέπει να υπάρχει λοιπόν η διαδρομή αυτή που θα συνδέεται με μια ε, ένωση, ένα σύλλογο ε, τοπικού χαρακτήρα και όλα αυτά να συνηφαίνονται σε ένα ε, νομικό καθεστώς με μια νομική βάση, γενικές συνελεύσεις, ένα διοικητικό συμβούλιο, μια δημοκρατικού χαρακτήρα διεργασία διαχείρισης ώστε μέσα σε ένα πλαίσιο κράτους δικαίου, μέσα σε αυτό το οργανικό πλαίσιο να μπορούν με δημοκρατικό τρόπο να διακυβερνώνται ή να αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης αυτη η διαδρομη ε, Θα πρέπει να υπάρχει και η αναγκαία ε, συνεισφορά και πρέπει να ε, συνεμπλέκονται τρεις χώρες, ένα άλλο κριτήριο το οποίο είναι σημαντικό, να συμμετέχουν τρεις χώρες κατελάχιστον σε τέτοιου είδους πολιτισμικές διαδρομές. Συνήθως συμμετέχουν περισσότερες χώρες αλλά το ελάχιστο, η ελάχιστη απέτηση από πλευράς κριτηρίων είναι η συμμετοχή τριών κρατών. Έχουμε 33 τέτοιες διαδρομές, 33 ε, όσον αφορά 57 χώρες. Έχουμε ένα ευρύτερο φάσμα λοιπόν γεωγραφικά ξεπερνάμε τα σύνορα, εντάσσεται το σύνολο της Ευρώπης και πέρα από αυτήν έχουμε κάποιες διαδρομές όπως την ε, διαδρομή των Βικίνγκων, ε, την, ε, τις διαδρομές του Ίνου για παράδειγμα που έχουν ένα ευρύτερο πλαίσιο συμμετοχής και πέρα από το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θρησκευτικές διαδρομές διασυνοριακές το πλαίσιο, το εύρος αυτού του προγράμματος είναι ευρύτατο λοιπόν, σε ένα πολύ ευρύ φάσμα. Έχουμε αρκετά παραδείγματα που θα θέλαμε να σας δώσουμε για να δώσουμε να αποκτήσει σάρκα και ωστά η εικόνα του τι βρίσκεται πίσω από αυτή την παρουσίαση. Θα ήθελα σύντομα να σας παρουσιάσω αυτή την πτυχή. Μερικά μονοπάτια για τα οποία έτσι αλλιώς περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στον ιστότοπο του Συμβουλίου. Έχουμε μοιράσει και ένα φυλάδιο που συνοψίζει τα πάντα και υπάρχει, υπάρχουν τα link για, στο website. Εδώ βλέπετε λοιπόν διάφορα τα μονοπάτια μας, αλλά υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες. Μιας λογής είναι αυτά που έχουν να κάνουν με το έδαφος. Οι διαδρομές λοιπόν κάποιες φορές έχουν να κάνουν ακριβώς με τη γη και τη χρήση της. Άλλη περίπτωση τέτοιων διαδρομών είναι αυτές των, ε, των αμπελιών ή των ελαιώνων στην Ανταλουσία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο. Άλλες είναι πιο γραμμικές διαδρομές. Ένα περιβόητο παράδειγμα η Via Francigena, η οποία είναι μια ε, διαδρομή που αφορά ένα κομμάτι, μια ζώνη που μπορεί κανείς να την περπατήσει κιόλα, κανονικά. Κάτι σαν την, ε, το προσκύνημα στον ε, Σαντιεγάγκο Ντακομποστέλα. Εδώ λοιπόν έχουμε τον βιώσιμο τουρισμό, τον αγροτουρισμό και προσκυνήματα τέτοιου τύπου όπως του Αγίου Ιακώβου. Επίσης υπάρχει η περίπτωση των δικτύων. Ένα από, μια από τις διαδρομές μας αυτές είναι αυτή του Μότσαρτ. Ένας δρόμος που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, απλώς μιλάμε για ένα σύμπλεγμα πόλεων με σημείων όπου ταξίδεψε, έζησε ο Μότσαρτ και είναι πραγματικά αξιοσημείωτη διότι 10 χώρες συνεργάζονται για αυτήν. Υπάρχουν τοπικές οργανώσεις σε αυτές τις χώρες που έχουν συνασπιστεί σε ευρωπαϊκή ομάδα των δρόμων του Μότσαρτ και κάνουν πολύ εντατική δουλειά με ένα πρόγραμμα πολύ φιλόδοξο. Πολλές δραστηριότητε, συναυλίες, αλλά και τέχνη αρχιτεκτονική που έχει να κάνει με τη ζωή του Μότσαρτ. Μετά έχουμε τα δίκτυα. Δίκτυα δρόμων. Αυτό είναι ακόμα ένα σύμπλεγμα διαφορετικών οδών, αλλά με διαφορετικές χώρες, διαφορετικά θέματα και κάποιες φορε διαφορετικε ιστορικε περιόδους. Πάντως υπάρχει κάτι κοινό, ένα ευρωπαϊκό στοιχείο πάντοτε σε αυτά. 25 ε, χώρες Εδώ η πόλη με κάστρα λοιπόν είναι ένα παράδειγμα ε, οι πόλεις με κάστρα και τύχη όπως ε, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, Και βλέπουμε την ιστορία κοινοτήτων ε, και ομάδων πληθυσμού και το πώς ζούσαν σε προηγούμενους αιώνες. Ένα από τα κριτήρια επιλογής στο οποίο επικεντρωνόμαστε έχει να κάνει και με την έρευνα. Ένα γνωστό παράδειγμα είναι πάλι η πολιτιστική διαδρομή του Κλουνί στη Βουργουνδία, στη Γαλλία όπου συμμετέχουν 11 χώρες που έχουν να κάνουν το αβαΐο Εδώ υπάρχουν εγκυκλοπαιδικά στοιχεία, υπάρχει η αποκατάσταση της ιστορικής εξέλιξης, είναι μια διαδρομή στην οποία μπορεί να περπατήσει πάλι κανείς κανονικά, αλλά υπάρχουν και πολιτικά στυλά που έχουν γίνει σε επίπεδο διαδικτυακό, ώστε οι Ευρωπαίοι από κάθε γωνιά να μπορούν να υποφεληθούν από αυτές τις ψηφιακές διαδρομές. Πολλές πληροφορίες λοιπόν διατηρούνται σε πλατφόρμες που ε, έχουν να κάνουν με τρεις διάστατες απεικονίσεις, ε, στοιχεία του αδαίου του κλουνί, το πώς έμοιαζε στο παρελθόν το Αδαΐο πώς εξελίχθηκε. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα Εδώ μια πτυχή που έχει να κάνει με τους νέους. Η τρανσρομάνικα, όπως έχει ονομαστεί οδός, με, το πολιτιστικό, με την πολιτιστική κληρονομιά της ρωμανικής περίοδου, που φέρνει κοντά πολλές διαφορετικές χώρες, όπου συμμετέχουν διαφορετικές συμμετέχουν νέοι από διαφορετικές χώρες, με πολλά ψηφιακά στοιχεία επίσης, Ε, που έχει να κάνει και με τις επισκέψεις μνημείων κάποιες φορές και σε ψηφιακό επίπεδο. Επίσης η οικονομική πτυχή είναι σημαντική διότι υπάρχουν και πολλές επιχειρήσεις που συνδέονται με αυτές τις οδούς πολλά προγράμματα επίσης που έχουν και οικονομική διάσταση όπως αυτή η οδός των ελαιώνων είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα με τοπικά προϊόντα τα οποία και χρησιμοποιούνται και προβάλλονται και η καλλιέργεια των ε, ελαιόδεντρων και η όλη κουλτούρα που την περιβάλλει παρουσιάζεται σε όσους ασχολούνται με αυτήν την οδό. Όπως είπα λοιπόν υπάρχουν κάποιες διαδρομές που μπορεί κανείς να τις περπατήσει στην Ευρώπη και στα μονοπάτια της. Η ο δρόμος του, του Αγίου Όλαφ είναι ένα παράδειγμα. για να γνωρίσει κανείς καλύτερα τις βόρειες περιοχές της Ευρώπης. Και επίσης ε, το προσκύνημα του Και ο Άγιος Ιάκωβος της Κομποστέλα είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. όπου βλέπουμε να συνδυάζεται η διαδρομή με την προσέλευση πολλών προσκυνητών ούτως ή άλλως. Όλα εξαρτάται βεβαίως από την ε, διάρκεια της διαμονής τους. Ε, είναι ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα, από τα πιο χαρακτηριστικά. Δεν είναι όλες οι οδοί τόσο πολύ σύχναστες, αλλά είναι ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα. Για να ολοκληρώσω λοιπόν να πω γιατί προσεκλήθη για να σας κάνω αυτή την παρουσίαση και να πω ότι σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας, ε, την Επιτροπή σας και για την εκπόνηση της έκθεσής σας το 2010 για τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Πολιτιστικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου και διεθνείς οργανισμούς καθώς και το γεγονός ότι έχετε προβλέψει συγκεκριμένα κονδύλια για συγκεκριμένα προγράμματα στον πολιτιστικό τομέα με ιδιαίτερη προσοχή στους ε, πολιτιστικούς δρόμους και μάλιστα αυτούς του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ευχαριστούμε λοιπόν για τη στήριξή σας. Έχουμε συνεργαστεί με την Επιτροπή για να μεταφράσουμε σε πράξη το ενδιαφέρον σας και να προωθήσουμε το ιδεώδες αυτό του να φέρουμε κοντά τους ανθρώπους από όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο μέσω του πολιτισμού με ένα θέμα κοινών ενδιαφέροντας, με έναν τρόπο που να είναι και βιώσιμος. Διότι όλοι αυτοί όλες αυτές οι διαδρομές είναι κάτι το μόνιμο. Είναι μία ομαδοποίηση τοπικών ε, ομάδων του πληθυσμού που στην πράξη συνδέονται και που μπορεί να έχουν κάποια χρηματοδότηση από τι αρχέ τοπική αυτοδιοίκηση, τι εθνικέ αρχέ ή τι ευρωπαϊκέ. Είναι λοιπόν ένα πολύ καλό μοντέλο γιατί είναι ακριβώ βιώσιμο. Η χρηματοδότηση πηγαίνει στου ανθρώπου στην πράξη. Το Συμβούλιο τη Ευρώπη έχει δικό του προπολογισμό που τροφοδοτείται από τα κάτι μέλη. Έχουμε ε, λοιπόν και υποχρέωση απέναντι στην Επιτροπή να προβάλλουμε την, ε, και να διαφημίσουμε αυτές τις διαδρομές, αλλά έχουμε και αυτές κάποια οικονομική δραστηριότητα. Το 2010 λοιπόν το Κοινοβούλιο δέχτηκε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πολιτιστικές διαδρομές και συνεργαζόμαστε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό μια σειρά από πρωτοβουλίες να αναφέρω ότι μια σειρά από διαδρομές έχουν αποφεληθεί από αυτή τη χρηματοδότηση απευθείας και αυτό είναι πολύ όμορφο διότι η πιστοποίηση του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι σαν ένα σήμα ποιότητας και μια εγγύηση ε, για την αξία των διαδρομών αυτών και την στήριξη της οποίας έτυχαν. Προκειμένου να παραμείνουν ζωντανές. Είναι λοιπόν σημαντικό να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε αυτό το επίπεδο, διότι το Κοινοβούλιο έχει όντω εντοπίσει συγκεκριμένα κονδύλια για αυτέ τι πολιτικέ διαδρομέ και ε, όντω το Συμβούλιο τη Ευρώπη κάνει διάκριση μεταξύ επιστοποίηση και με επιστοποίηση. Η τελευταία μου διαφάνεια αφορά τα προγράμματα που μπορέσαμε μαζί με τη δική σας στήριξη και της Επιτροπής της DG Grow σε μια σειρά ετών να ε, αναπτύξουμε. Τα προβάλαμε τουλάχιστον ε, τα προγράμματα και τις διαδρομές με τρόπο ώστε να ωφελήσουμε το δίκτυο, να διευρυνθεί, να προσελκύσουμε ενδιαφέρον υποψηφίων, υποψηφίου που μπορεί να ζητούν πληροφορίε, δεν ξέρουν ακριβώ πώ να τα σχεδιάσουν όλα αυτά. Είχαμε λοιπόν πολλέ αιτήσει για πιστοποίηση. Όλα αυτά επιτρέπουν στο Συμβούλιο τη Ευρώπη να προωθήσει το πρόγραμμα αυτό. Έχουμε ρόλο συντονιστή, αλλά πραγματικά την ε, πραγματική ευθύνη την έχουν οι ίδιοι οι διαχειριστές του προγράμματος. Σας ευχαριστώ πολύ και αναμένω τη συζήτηση μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Θα συνεχίσω στα τελικά για τα τελευταία σχόλια να πω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αυτό είναι ένα πρόγραμμα πραγματικά συναρπαστικό και συνεχίζει να είναι. Μας δώσατε κάποια δεδομένα. Είπατε για τον Άγιο Ιάκωβο της Κομποστέλα. Αλλά και για την ε, Φραντίντζενα... αυτήν την οδό, που βλέπουμε να επισκέπτονται τόσες χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο. Τώρα για τις διαδρομές του Σαντιάγκο λόγου χάρη και ε, την ε, διαφραγγική οδό. Πολλές φορές ακούμε ότι οι διαδρομές ε, μπορεί να συζητώνται από εμά, αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί που τις περπατάμε. Εγώ πρέπει να πω ότι σε μια από αυτές τις διαδρομές πήγα και περπάτησα και ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστες εμπειρίες, θαυμάσιες μάλλον εμπειρίες και αυτή του Αγίου Ιακώβου της Κομποστέλα και τη, η διαφραγική οδός. Εδώ λοιπόν πρέπει να πλευρεύσουμε μια γραμμή προπολογισμού, ακόμη και μικρούτσικη για να στηρίξουμε αυτά που πρότεινε το Κοινοβούλιο. Μια νέα γραμμή λοιπόν του προπολογισμού σε ό,τι αφορά τον βιώσιμο πολιτιστικό τουρισμό. Εδώ αίτηση θα πρέπει να μπορούν να ε, υποβάλλουν και οι υπεύθυνοι διαδρομών και οι πιστοποιημένες διαδροπές βέβαια αλλά και οι νέες θέλαμε να υπάρχει μια σχετική ισορροπία μεταξύ των δύο, κατηγοριών. Τώρα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Ποιος θέλει. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να με συγχωρήστε που είμαι σε τέτοια υπερδιέγερση σήμερα το πρωί, αλλά τα θέματα στην ημερήσια διάταξη με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Να σας ευχαριστήσω δε για την παρουσίαση που κάνατε. Και πρέπει να σας πω πως οι διαδρομές είναι πολύ σημαντικές και το λέω ως πρώτο. Ξέρετε πως ε, ξεκάθαρα οι διαδρομές αυτές χαρακτηρίζονται από τον όρο Ισπανία. Και είναι πολύ δύσκολο να βρούμε μία από αυτές τις διαδρομές οι οποίες να μην ε, ε, αποτελούνται από ένα τμήμα ισπανικό. Για ποιο λόγο έχουμε αυτή την ισπανική κυριαρχία. Είναι θέμα ιστορικό αυτών των διαδρομών ή υπάρχει κάποιος άλλος για τον οποίο έχουν τόσο διακριτό ρόλο οι Ισπανοί. Και επίσης οργανώνεται διασκέψεις, για παράδειγμα συναισθιάσεις, ε, ημερίδες για όσους τρέχουν αυτές τις διαδρομές έτσι ώστε να ανταλλάσσουν εκεί τις βέλτιστες πρακτικές. Επίσης, τα νεκροταφεία. Έχω δει πως υπάρχει ε, μία σειρά από πολύ ενδιαφέροντες τόπους νεκροταφείων Οπότε, ε, είμαι πολύ ικανοποιημένο, αλλά λείπει το Auschwitz-Birkenau, το οποίο είναι ένα μεγάλο νεκροταφείο και αν δεν τοποθετήθηκε στη διαδρομή των νεκροταφείων, ε, θα ήθελα να με εξηγήσετε για ποιο λόγο, γιατί όντως αποτελεί κομμάτι της ε, κληρονομιάς μας. Επίσης, κοίταξα και τη διαδρομή της ε, Ιουδαϊκής ε, ε, πολιτιστικής κληρονομιάς. Πολύ ε, καλή η περιγραφή, αλλά λείπει από το κομμάτι αυτό η Πολωνία. Ε, και εμεί είχαμε ένα μεγάλο κομμάτι ε, εβραϊκού πληθυσμού και δεν βλέπω να εμφανιζόμαστε. Επίσης έχουμε και τη διαδρομή με τα πάρκα και τους κήπους. Πολύ η διαδρομή και αυτή. Γιατί όμως δεν έχουμε καθόλου ιαπωνικού τύπου κήπων ε, σε αυτή τη διαδρομή, γιατί υπάρχουν πολλοί εξαιρετικοί τέτοιοι κήποι στην Ευρώπη. Υπάρχει τρόπος να προσθέσουμε ε, κάποια σημεία στις διαδρομές αυτές. Και βέβαια είναι πολύ καλό που κάνετε εσείς τον ποιοτικό έλεγχο και που πιστοποιείτε αυτές τις διαδρομές. Θα ήθελα να ε, σας από για το γεγονός ότι πιστοποιείται έτσι ώστε να υπαλληθεύεται κάπως πως οι διαδρομές αυτές εξακολουθούν να αξίζουν αυτό το χαρακτήρα το χαρακτηρισμό μάλλον και θα ήθελα να πείτε τέλος πώς γνωρίζουμε εάν έχουν κατατεθεί νέες αιτήσει πιστοποίησης πώς μπορώ να ξέρω εγώ για παράδειγμα αν κάποιος ε, υπέβαλε αίτηση που βρίσκεται η αίτηση αυτή και πόσο χρόνο χρειάζεται ε, ποια είναι η πιο σύντομη προθεσμία για μια αίτηση να εγκριθεί Προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον η παρουσία σας και πάρα πολλοί θέλουν το λόγο. Η κυρία Τρούπελ. Yes, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Κάνατε λόγο για το ότι είναι σημαντικό στο επίπεδο των πολιτών οι ιδέες αυτές ε, να μπορούν να βρίσκουν την αποδοχή τους και να εφαρμόζονται. Αλλά θα πρέπει να δούμε πώς αυτό θα μπορεί να γίνει διαφημίζοντας το ή ενθαρρύνοντας και προτρέποντας ε, τους πολίτες ε, να εμπλακούν και να δράσουν σε αυτό το πλαίσιο. Ευχαριστώ. Άλλοι που θα ήθελα να παρέμβουν. Μαραγκάζω παρακαλώ. Μπορώ να μιλήσω ισπανικά. Μπορώ να μιλήσω ισπανικά. Μπορώ να μιλήσω και ιταλικά αν θέλω. Mm. Εν πάση περιπτώσει, ακούγοντάς αυτό το πρόγραμμα πραγματικά θα μπορούσε να δώσει πολλά περισσότερα και να απαιτήσει κανείς ε, υπό το έννοια ε, βελτίωσης όχι σε σχέση με το σχέδιο ή το περιεχόμενο αλλά για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε περισσότερο σε στόχους σημερινούς και ανησυχίες ε, στην Ευρώπη σημερινές επικαιροποιημένες. Ο καλύτερος τρόπος ε, που θα μπορούσε να ε, γίνει αυτό και να κατανοήσει κανείς αυτές τις αλλαγές είναι να δει κανείς ε, το ιστορικό πλαίσιο και να κατανοήσει το ιστορικό πλαίσιο. Χωρίς αυτό βλέπει κανείς μνημεία, καλλιτεχνικά δημιουργήματα Υπάρχει όμως μια αξία στην, στο σημερινό πλαίσιο που θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη επίπτωση όλα οι διαδρομές που συσχετίζονται με την παρουσία διαφορετικών πολιτισμών για παράδειγμα ένα σαφές παράδειγμα την παρουσία της Τουρκίας για παράδειγμα στην κεντρική Ευρώπη ένα παράδειγμα αναφέρω ή την αξία της ε, ενιαίας ε, ας το πω έτσι της διάστασης των ευρωπαϊκών πόλεων της διάστασης των πόλεων πόλης ως ε, μια καλύτερη αποκριστάλλωση του τι είναι η Ευρώπη. Η Ιταλία είναι ένα υποδειγματικό τέτοιο παράδειγμα με τις πόλεις ε, κράτης, κράτη και με την, ε, τον ρόλο τους στην δημιουργία και αποκριστάλλωση της Ευρώπης ιστορικά. Σοντρόβα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα να επικεντρωθούμε λίγο περισσότερο στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης σε σχέση με τα πολιτικά δικαιώματα και δικαιώματα του ανθρώπου. Αυτό είναι ο λόγος ύπαρξης εξάλλου του Συμβουλίου της Ευρώπης ο πολιτισμός είναι μια πολύ σημαντική διάσταση και έχει τεράστια σπουδαιότητα για το Συμβούλιο της Ευρώπης και συνεργάζεται σε σχέση με τα θέματα πολιτισμού και παιδείας και εκπαίδευσης ε, το Συμβούλιο της Ευρώπης και ελπίζω ότι θα συνεχίσει αυτή η δραστηριότητα και θα ανθίσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η συμμετοχή και να εποφεληθούμε από την πραγματογνωμοσύνη και γνώση γνώση που έχει το Συμβούλιο της Ευρώπης όσον αφορά την παιδεία και την εκπαίδευση. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω ποιες είναι οι εμπειρίες σας, ποια, τι, τι είδατε σε σχέση με την δημοκρατία της Τσεχίας. Υπάρχει ίσως κάποιο πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει η Τσεχία. Ευχαριστώ πολύ για το έργο που επιτελεί. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της χρηματοδότησης αν επιτρέπετε ποια μορφή παίρνει μακροπρόθεσμα η χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων και σχεδίων. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι που από πλευράς περιεχομένου ε, έχουμε προκατακτικές δράσεις, ε, απαιτείται ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ώστε να μπορέσει να τύχει χρηματοδότησης. Ήδη το έργο που έχει επιτελεστεί για παράδειγμα θα με ενδιαφέρε μακροπρόθεσμα να μου πείτε πώς θα μπορούσαν τέτοια προγράμματα να είναι, ας το πω έτσι, να μπορούν να καλύπτουν τα έξοδά τους και να είναι ε, τα πιο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Ναι, αλλά πραγματικά σημασία έχει και πώς οι ενώσεις των πολιτών, οι ομάδες τους και οι σύλλογοι, δηλαδή από κάτω προς τα πάνω, μπορεί να επιτρέψει διαπολιτιστικό διάλογο. Ξέρω δύο παραδείγματα, να τα αναπτύξω. Η φραγκογενής οδός όπως ονομάστηκε που αφορά τέσσερις χώρες και πάρα πολλές ε, τοπικές κοινότητες έχει φτιαχτεί από μια ομάδα κοινοτήτων της φραγκογενούς οδού που μαζί από, με τις σχετικές ενώσεις ε, την ε, στηρίζουν και ευαισθητοποιούν για παράδειγμα τις διάφορες επαρχίες για το πόσο πρέπει να προβλεφθούν πρωτοβουλίες αλλά και να δαπανηθούν ε, συγκεκριμένα κονδύλια μέσω των διαφορετικών ταμείων και το λέω γιατί το ξέρω εκ πείρας. Όπως υπάρχει το Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ της ε, Φραγκογενούς Οδού ε, το οποίο το ε, πλαισιώνουν, το κινούν ουσιαστικά οι καλλιτέχνες οι ίδιοι, η μουσική με μουσική μεσαιωνική σε όλες τις περιοχές της οδού αυτής κάτι που επιτρέπει να τροφοδοτηθεί η όλη προσπάθεια και να πω και ένα άλλο παράδειγμα γιατί η διακυβέρνηση από κάτω προς τα πάνω είναι κάτι που το έχω ζήσει στην πράξη. Δεν είναι εύκολο, αλλά και σε άλλες οδούς συμβαίνει αυτό. Κάποιοι έχουν πετύχει περισσότερα, κάποιοι λιγότερα, αλλά κάποιοι έχουν πετύχει ακόμη και να εμπλέξουν τα πανεπιστήμια στην έρευνα της ιστορίας, όχι μόνο των μνημείων και των αξιοθεάτων, αλλά για τις συναντήσεις, την ιστορική διαστρωμάτωση, Υπάρχει διεύρυνση της συμμετοχής από θεσμού ενώσεις και συλλόγους μέχρι ομάδες πολιτών. Το βρίσκω μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κώστα να επιβεβαιώσω αυτό που μόλις είπατε ότι η ομορφιά του προγράμματος είναι πως κάθε διαδρομή έχει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δραστηριότητα. Δεν είναι μόνο εθνικό, τοπικό, περιφερειακό, το οποίο μοιράζεται και κατακαιρματίζεται μεταξύ διαφορετικών πραγματικότητων. Όχι, η ευρωπαϊκή διάσταση υπάρχει σε όλες τις ε, διαδρομές. Οπότε κάθε χρόνο παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο είναι ευρωπαϊκό και καλούν μέλη από τις άλλες χώρες, ε, εκ περιτροπής αν ε, αλλάζουν τον χώρο στον οποίο συναντιέται η Ένωση έτσι ώστε να υπάρχει μια γονιμοποίηση των ιδεών άρα δεν μιλάμε για εθνικά προγράμματα γιατί αυτές οι πολιτικές διαδρομές είναι ουσιαστικά ομοσπονδίες χωρών και αυτή είναι και η ομορφιά τους δηλαδή συναντιόνται σε ένα κοινό θέμα για παράδειγμα, είναι η γραμμή της αγιοπλαστικής, η διαδρομή της αγιοπλαστικής που έχουμε κεραμιστές από πολλές χώρες που μοιράζονται το πάθος τους ε, κατά καιρούς. Χαίρομαι γιατί θίξατε πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Η πρώτη είναι αυτή που μας έκανε ο Πολωνός συνάδελφός σας, γιατί ήταν πολύ σχετικές οι παρατηρήσεις του για τις βέλτιστες πρακτικές και τις ε, συνεδριάσεις και τα συμπόσια και τις ε, συνδιασκέψεις, ό,τι μπορούμε με τον περιορισμένο προϋπολογισμό που έχουμε. Αλλά μέσα στη χρονιά μια σειρά εκδηλώσεων λαμβάνουν χώρα όπου εκπαιδεύουμε τους διαχειριστές αυτών των πολιτιστικών διαδρομών είτε στο Στρασβούργο είτε στο Λουξεμβούργο και καμιά φορά σε κάποια από διαδρομές όλους μαζί, όλους τους 33 λοιπόν διαχειριστές και πολλές φορές εκπροσωπούνται με παραπάνω από ένα άτομο από κάθε δερμή, όπως επίσης και του υποψηφίου που χρειάζονται να πιστοποιηθούν, οπότε συνήθω έχουμε γύρω στα 50 άτομα και παραπάνω και του εκπαιδεύουμε. Δεν είναι ακριβώς εκπαίδευση, είναι μια ανταλλαγή πρακτικών, γιατί πρέπει να κατανοήσετε πω η πιο παλιά πολιτιστική διαδρομή είναι του 87 και έχουμε και κάποιες οι οποίες γεννήθηκαν τα δεκαετία του 90, του 2000, του 2010, πέρσι εγκρίναμε και προσωπήσαμε και άλλες. Έχουμε νέες διαδρομές που είναι πιο νέες. Έχουν λιγότερη εμπειρία στη διαχείριση και ε, στην κοστολόγηση και τους ε, ε, φέρνουμε σε επαφή και με τα πανεπιστήμια, γιατί έχουμε και δίκτυο πανεπιστημίων. Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, αρκετά πανεπιστήμια όπου έχουμε προγράμματα μάστερς για την πολιτιστική κληρονομιά και στηρίζουν ως πραγματογνώμονες για το πώς μπορεί να διαχειριστεί κανείς ε, τέτοιου είδους διαδρομή και τους ε, προσφέρουμε ένα τόπο ανταλλαγής ε, απόψεων μεταξύ υποψηφίων αλλά και επιστοποιημένων διαδρομών και πολλές φορές Έχουμε θεματικές ιδέες όπως για παράδειγμα τι σημαίνει η ιδέα της Ευρώπης. Πέρσι, για να σας πω, Μιλήσαμε για τη δικτύωση. Ε, φέτος θα μιλήσουμε για την εμπορική προώθηση ως πολιτικό, ως τουριστικό με συγχωρείτε προϊόν. Εσείς μιλήσατε και για το θέμα του γιατί η Ισπανία έχει τόσες διαδρομές, γιατί η Πολωνία δεν έχει τόσες φαντάζομαι. Η δημοκρατική ομορφιά αυτών των διαδρομών είναι πως είναι οι ίδιες οι χώρες οι οποίες καταθέτουν τις προθέσεις τους ε, και ζητούν να ε, λάβουν μέρος σε συγκεκριμένη διαδρομή. Εμείς δεν υποχρεώνουμε κάποιον, δεν λέμε στην Πολωνία η Πολωνία πρέπει να γίνεις μέλος. Είναι δημοκρατική η διαδικασία και αν κάποια χώρα σε τοπικό επίπεδο και μέσω Υπουργείων θέλουν να συνδεθούν με μια συγκεκριμένη διαδρομή γιατί υπάρχει μια τοπική δραστήρια κοινότητα που ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό, για την ιστορική περίοδο, για την αρχιτεκτονική, για οτιδήποτε μέσω της Ένωσης συνδέεται και το Συμβούλιο της Ευρώπης πιστοποιεί τη διαδρομή βασιζόμενο στα ε, κριτήρια τα οποία σας περιέγραψα αλλά αφήνει τη διαδρομή να αναπνεύσει. Έχει τη δική της ζωή και μπορεί να είναι μια μεγάλη διαδρομή. Έχουμε διαδρομές με 15 χώρες, 20 και άλλες είναι πιο μικρές. Γιατί το ίδιο το θέμα δεν μπορεί να επεκταθεί πολύ. Για παράδειγμα, κάποιες διαδρομές δεν μπορούν να περάσουν de facto πάνω από 5-6 χώρες γιατί είναι μια κοινή ιστορική ε, ταυτότητα. Για παράδειγμα, η διαδρομή του Ναπολέοντα. Ε, εντάξει, αυτό θα καλύψει μόνο εκεί που έζησε ε, και πολέμησε. Ή κάποια χώρα που έχει μουσείο του Ναπολέοντα, αλλά είναι σχετικά περιορισμένο. Μότσαρτ είναι περιορισμένος ο αριθμός χαρών, ο οποίος επί της αρχής μπορούν να, να ε, συνδεθούν. Οπότε θα πρέπει καταρχήν οι χώρες να εκφράσουν την επιθυμία και μετά η Ένωση έχει την υποχρέωση να υποδεχτεί τα νέα μέτρα και αυτό γίνεται και σε επίπεδο εργανώσεων βάσης που είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν είναι μια, ε, ένα πρόγραμμα το οποίο επιβάλλεται από την κορυφή προς τη βάση αλλά ε, ξεπηδά από την ίδια τη βάση. Άλλοι χώρες ενδιαφέρονται περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Αλλά επειδή έχω αναλάβει τη διεύθυνση αυτού του προγράμματο, θέλω να σα πω πω στόχο μου είναι στην Ανατολική Ευρώπη και στην Νότια Ανατολική Ευρώπη να επεκτείνουμε. Γιατί γεννήθηκε την 70 και το 80 το πρόγραμμα αυτό και υπάρχει μία στροφή προς τη Δυτική Ευρώπη η οποία υπερεκπροσωπείται. Και το Συμβουλίο της Ευρώπης όντως φέρει κάποια ευθύνη, είμαστε 47 μέλη, οπότε θα πρέπει να καλύψουμε όλη την Ήπειρο. Ε, ε, not... Θα πρέπει λοιπόν να καλύψουμε και χώρες οι οποίες δεν εκπροσωπούν ιδιαίτερα, να μιλήσουμε εκεί με τις τοπικές κοινωνίες και τις αρχές. Ο διευθυντής μου είτε αυτή την εβδομάδα την επόμενη πάει στη Βαρσοβία για να μιλήσει με το Υπουργείο ε, Πολιτισμού. Γενικώ γιατί θα πάει στη Μόσχα για να μιλήσει με τη Ρωσική Ομοσπονδία. New countries and new Με νέε διαδρομέ. Νέε διαδρομέ. Γιατί μέχρι σήμερα η στρατηγική μα ήταν και έτσι το κάναμε στο παρελθόν να περιμένουμε εμεί να μας καταθέσουν τις αιτήσει. Να περιμένουμε εμείς να ενδιαφερθούν. Τώρα η προσέγγιση δική μου είναι λίγο διαφορετική, είναι πιο ενεργητική. Δηλαδή να πούμε ότι υπάρχει ένα, ένας θεματικός χώρος τον οποίο εμείς δεν εκπροσωπούμε. We solicit and we can help because we are... Πού μπορούμε να ζητήσουμε να συνδεθούν μαζί μας. Είμαστε πραγματογνώμονες. Έχουμε την τεχνογνωσία, για παράδειγμα. Υπάρχει μια διαδρομή που είναι ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος. Είναι πνευματικής η, η διάσταση αυτή η διαδρομή και υπάρχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί είναι ε, για συγκεκριμένο δόγμα. Οπότε μας αρέσει η ιδέα του να ε, έχουμε και τη διαδρομή του αλατιού για παράδειγμα όπου είχαμε την εξόριξη ή την Παρασκευή άλατος συγκεκριμένες κοινότητες που έχουν τεχνογνωσία. Είναι ένα σχέδιο και αυτό. Uh, Στην περιοχή της Βαλτικής έχουμε μια ένωση η οποία ε, προσπαθεί να συνδέσει και όλα τα κάστρα. Υπάρχει, υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά η διαφορά μεταξύ μιας υποψηφιότητας και μιας πιστοποιημένης ε, διαδρομής είναι η πολλή δουλειά που χωρίζει στις δύο. Οπότε ναι. Το πώς μπορεί κανείς να προσθεθεί σε μια διαδρομή, αν μια τοπική κοινότητα θέλει να γίνει μέλος, υπάρχει ένωση, υπάρχει διαχείριση και είναι εύκολο να γίνει κανείς μέλος. Και η ομορφιά του προγράμματος είναι, και νομίζω αυτή ήταν η ερώτηση της κυρίας Βεράιν για τη χρηματοδότηση, είναι που σε κάποιο βαθμό είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Έχουμε κάποιες διαδρομές που είναι διαδρομές 25-30 χρόνια. Όχι γιατί χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά γιατί υπάρχει συμμετοχή που στηρίζει οικονομικά τη διαδρομή. Και αυτό αποδεικνύει το ότι λειτουργεί το πρόγραμμα. Τον 1999 έχουμε τη Χανσιατική, έχουμε την ε, Φραγκογενή, έχουμε πάρα πολλές. Το 2002 το Μότσαρτ. Είναι βιώσιμα project, αυτό χρηματοδοτούμενα για αρκετά χρόνια και πολλές φορές βέβαια θα λάβουν συγκεκριμένη ε, επιδότηση χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν εξαρτώνται από αυτή την ε, χρηματοδότηση. Και αυτό είναι κάτι διαφορετικό από διαδρομές οι οποίες γεννώνται ως ε, project με χρηματοδότηση και μόλις διακοπεί η χρηματοδότηση εξαφανίζονται. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από αιτήσει, δεν τις κοιτάμε όλες. Τρία με πέντε χρόνια πάντως παίρνει η διαδικασία γιατί η νομική αρχιτεκτονική χρειάζεται δηλαδή η ένωση, η, τα μέλη, το νομικό πλαίσιο και αυτό δεν είναι πάντα τόσο εύκολο. have... Αλλά αυτό είναι που επιτρέπει ακριβώς τη βιωσιμότητα, να έχεις μια νομική οντότητα και μια επαφή με την τοπική κοινωνία, μια σχέση με αυτήν που σε προωθούν περισσότερο γιατί αποκτάς μια ε, πιο έντονη παρουσία. Η κυρία Τρούπελ με ρώτησε για το τι γίνεται με την εκπροσώπηση της βάσης και πώς μπορούμε εμείς να ε, απευθυνθούμε σε περισσότερους ανθρώπους. Έχει να κάνει με την ίδια τη διαδρομή, με το πώς διαχειρίζονται, με το πώς μπορούν να επεκταθούν ε, και εμείς βοηθάμε με κάποια στήριξη, αλλά η φύση του project είναι τέτοια που η ίδια η διαδρομή πρέπει να βγει έξω να βρει νέα μέλη. Και αν δείτε, πολύ συχνά έχουμε νέες χώρες, νέα σημεία και αυτά φαίνονται και από το χάρτη μας. Είδατε η Πολωνία και στην Πολωνία έχουμε αρκετές, αρκετούς δήμους. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια εξάπλωσης θα πρέπει να γίνει από την ίδια τη διαδρομή γιατί έχει τη δική της ζωή. Τώρα, για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα επικαιρότητα. Πολύ σημαντικό αυτό και για ιστορικούς λόγους και για να μπορούμε να ανατρέξουμε στην ιστορία μας. Είναι σημαντικό σήμερα να δούμε πώς μπορούμε να προσθέσουμε μια σειρά διαδρομών, να μιλήσουμε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι σε μεγάλο βαθμό πολιτιστικό project, αλλά παράλληλα είναι και πολιτικό project. Δηλαδή, δημοκρατικό, αλλά project παρόλα αυτά, που δείχνει ποιες είναι οι προκλήσεις της σημερινής Ευρώπης. Εμείς προσπαθούμε να συνεισφέρουμε στις προκλήσεις αυτές, δείχνοντας πως μαζί θα σταθούμε, μοιραζόμαστε μία κοινή ταυτότητα η οποία μας ενώνει περισσότερο από ό,τι μας χωρίζει και η ομορφιά είναι ότι μπορεί να βρει κανείς θέματα τα οποία ενδιαφέρουν όλους τους Ευρωπαίους. Γιατί τελικά είναι τόσα πολλά τα κοινά μας στοιχεία. Σε πνευματικό επίπεδο, σε πολιτισμό, σε τέχνη, σε πολλά. Οπότε προσπαθούμε όσο μπορούμε. Κύριε Στυροβα, ήθελα να σας πω πως υπάρχει και το θέμα της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Εμείς αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτή τη συνεργασία και θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και το λέμε συχνά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει μέλος. Κατανοώ πως υπάρχουν κάποια νομικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να mm. ε, εξεταστούν, αλλά νομίζω πως θα μπορούσε να γίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση κομμάτι του σώματος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χάρη στη δική σας ε, ε, γραμμή του προπολογισμού που έχει δοθεί στις πολιτικές διαδρομές έχουμε πετύχει ένα υψηλό επίπεδο συνεργασίας που θα θέλαμε να συνεχιστεί. Νομίζω η Τσεχία θα μπορούσε να κάνει παραπάνω για να αναπτύξει τέτοιου είδους πολιτιστικές διαδρομές. Πάντως, θα μπορούσαν ίσως να γίνουν μέλη με την Τσεχία θα θέλαμε να συνεργαστούμε ως χώρα και ως πολιτισμός και πολιτικό κέντρο έχει τόσα να προσφέρει. Οπότε είναι κρίμα που δεν είναι πιο δραστήριο. Οπότε προσπαθούμε εμείς να τα δούμε στο Στρασβούργο και βέβαια μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού. Γιατί εμείς χρειαζόμαστε τέτοιου είδους δέσμευση. Τέλος, Uh, I have Για τη χρηματοδότηση, κυρία Βερέν, να σας πω πως το πόσο βιώσιμα είναι όλα αυτά, νομίζω είναι αρκετά βιώσιμα. Είναι αυτοχρηματοδοτούμενα και ο μηχανισμός τους δίνει τη δυνατότητα να επιβιώνουν και να συνδέονται με το χώρο στον οποίο βρίσκονται. Και πολλές από αυτές τις ε, διαδρομές ε, λαμβάνουν και τέλη σε τοπικό επίπεδο από τις κοινότητες, από τους δήμους. Καλό είναι βέβαια να επεκτείνεται κανείς και αυτή η αυτοχρωματοδότηση πολλές φορές είναι περιορισμένη. Look at it in a broader perspective. One is the economic aspect of the routes. And then there is... Και βέβαια σε όλα αυτά θα πρέπει να δούμε και την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν οι διαδρομές στον ίδιο το χώρο στον οποίο βρίσκονται. Οι αριθμοί είναι πολύ μεγαλύτεροι από αυτό που φαίνεται στο χαρτί. Δηλαδή, όταν μιλάμε στο παραδοτέο, σε αυτό που προσφέρουμε, όταν κοιτάμε τις δίκτυα και τις διαδρομές, οι επιπτώσεις, για παράδειγμα, σε τουριστική καρποφορία, είναι πολύ υψηλές, γιατί υπάρχει προσθέμενη αξία της δικτύωσης και ένας πολιτιστικός περιηγητής, ένας τουρίστας θα πάει ένα χρόνο σε ένα κομμάτι της διαδρομής και μετά την επόμενη χρονιά θα πάει να ταξιδέψει ή να έχει την εμπειρία ενός άλλου κομματιού της διαδρομής. Να σας δώσω το παράδειγμα των ε, ιστορικών ιαματικών πόλεων. Ξέρετε πως υπάρχουν πολλές ιαματικές πόλεις ε, στην ε, Ευρώπη και τη μια χρονιά θα πάνε στη μια πόλη και επειδή μαθαίνουν ότι υπάρχει δίκτυο ολόκληρο θα επισκεφτούν μια επόμενη χώρα και ένα επόμενο κομμάτι την επόμενη χρονιά. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει αυτή η αίσθηση έτσι ώστε ο τουρίστας να επαναλάβει την εμπειρία αργότερα. Και έχουμε πολλές ιδέες πώς να γίνει αυτό. Υπάρχει ένας τρόπος λοιπόν σύνδεσης με τον τουρίστα έτσι ώστε να γίνεται πιστός φίλος της διαδρομής και να θέλει να επαναλάβει την εμπειρία σε κάποιο άλλο σημείο. Όπως επίσης και η βιωσιμότητα αυτές τις διαδρομές. Είδατε ότι υπάρχει το πρόβλημα της εποχικότητας. Η ομορφιά του προγράμματος είναι ότι πολλές από αυτές τις διαδρομές αφοφορούν όλη τη χρονιά. Και δεν νομίζω ότι μπορείς να περπατήσεις όλες τι διαδρομές το Δεκέμβριο. Δεν πάει κανεί στην Νορβηγία Λίμον, Δεκέμβριο, ούτε στη Σουηδία. Αλλά υπάρχει μία περίοδος ε, γόνιμη για όλες αυτές τις διαδρομές, τις οποίες μπορεί κανείς να απολαύσει για μία σειρά λόγων με πολλούς κονοσέρ όλων των ηλικιών. Μιλήσαμε για του νέου. Um, Έχουμε και τους ηλικιωμένους. Um, um, Εγώ για παράδειγμα πήγα σε μια παρουσίαση στο Λουξεμβούργο. Και μας είπαν μπορούμε να πάμε ως tour. Οργανωμένη δηλαδή εκδρομή. Και μου είπαν όχι δεν γίνεται. Τους είπαμε όχι δεν γίνεται. Αλλά αν σας ενδιαφέρει ο Μότσαρτ, μπορώ να σας φέρω σε επαφή για να κάνετε κάτι αντίστοιχο, να κάνετε ένα τούρ. Και πρέπει να σας πω πως ο πολιτισμός, το ξέρετε, είστε η Επιτροπή Πολιτισμού, είναι θησαυρό για την Ευρώπη, με εξαιρετικά υψηλή αξία και ένα από τα στοιχεία που εξασφαλίζει το οικονομικό μέλλον της Υπήρου μας είναι η διατήρηση ε, και η ανάδειξη του πολιτισμού και της πολιτιστικής μας ε, κληρονομιάς. Η Ευρώπη είναι πανέμορφη και θα πρέπει να την αναδείξουμε μια και υπάρχει το δυναμικό να την απολαύσουν όχι μόνο οι Ευρωπαίοι αλλά και οι μη Ευρωπαίοι. Ε, through these cultural is also uh, service and και γι' αυτό πρέπει να σου πω ότι δεν έχουμε μόνο τους παραδοσιακούς προορισμούς και αυτό πρέπει να το πούμε απερίφραστα. Εντάξει Βενετία, εντάξει η Ρώμη, εντάξει το Παρίσι, ε, εντάξει η Πράγα. Αλλά υπάρχει και το υπόλοιπο. Ωραία, έχουμε τους πύργους στη Γαλλία, του Λίγυρα. Είναι λίγα, πάνε πολύ, 20 χιλιόμετρα γύρω από το Λίγυρα από, μακριά από τη, ε, τους πύργους αυτούς δεν πάει κανείς γιατί δεν τα ξέρει. Λοιπόν, υπάρχει μια όμορφη Ευρώπη που έχουμε στη διάθεσή μας. Και υπάρχει μια προστιθέμενη αξία η οποία είναι και πολύ δημοκρατική. Και βέβαια με την εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών. Γιατί με τον τρόπο αυτό θα εμπλουτίσουν την οικονομία τους και βεβαίως υπάρχει και ο μικρός ρόλος που είναι, για παράδειγμα, η διαδρομή του Στίβενσον που περνάει από τη Γαλλία, έρχεται από την Αγγλία μέσω Βελγίου στη Γαλλία και είναι η διαδρομή που έκανε ο Στίβενσον, ο συγγραφέας, όσο έγραφε τα βιβλία του για τον νησί των θησαυρών κτλ. Και έρχομαι και τώρα από ε, που, που, από την Αμερική γιατί έρχονται οι Αμερικάνοι να δούνε πού έζησε, πού έγραψε αυτός ο άνθρωπος και αυτό βέβαια εξυπηρετεί και την τοπική οικονομία, μια και συνεισφέρει και οικονομικά. Ξέρω πως είστε Επιτροπή Πολιτισμού. Αλλά ο πολιτισμός, εκτός από ο πολιτισμός, είναι και η οικονομία του πολιτισμού. Μην το ξεχνάμε, σας ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα, κύριε Ντομινιάννη, και για, για το πάθος σας, το ζήλο αυτό στη δουλειά σας. Είμαι βεβαία ότι αυτό το υπέροχο πρόγραμμα θα προχωρήσει ακόμα καλύτερα και στο μέλλον. Να χαιρετήσω και τον συνάδελφο Μίλαν διότι μαζί του εργαστήκαμε στην ε, διακομματική ομάδα για τα πολιτιστικά αθλητικά θέματα και την ψυχαγωγία. Ε, νομίζω ότι επειδή αναφέραμε τις δύο μεγάλες οδούς ε, του Αγίου Ιακώβου και την Φραγκογενή, έπρεπε να σας χαιρετήσω και εσάς γιατί είχατε συμμετάσχει ε, στις επισκέψεις και για την ε, διαπιστημονική σημασία του θέματος. Τώρα λοιπόν ας κλείσουμε λέγοντας ότι μας ενδιαφέρει βεβαίως ως Κοινοβούλιο να έχουμε και άλλες μορφές συνεργασίας μαζί σας, με το Συμβούλιο της Ευρώπης, με το Ινστιτούτο σας, για να είμαστε όχι απλώς ε, συμμέτοχοι της προσπάθειάς σας, αλλά και να στηρίξουμε περαιτέρω την προβολή του προγράμματος αυτού. Γίνεται πολύ λεγός για narrative, για αφήγημα, το νέο αφήγημα της Ευρώπης. Εδώ λοιπόν μην ξεχνάμε τι ε, ίχνη υπάρχουν στην Ευρώπη σε όλα αυτά τα μονοπάτια της ε, Ευρώπης αυτής. Μετά είναι και ο ρόλος των τοπικών κοινοτήτων που διαρκώς αυξάνεται. Ξεπερνώνται οι τοπικισμοί και δημιουργείται μια διαδρομή που μπορεί να ξεπερνά τα όρια μιας χώρας. Ε, συμμετέχουν και άλλες κοινότητες, οπότε ξεπερνάει κανείς τη μικρόνιά του. πρόκειται για ένα ευρωπαϊκής εμβέλειας εγχείρημα. Αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρξουν συγκεκριμένε προβλέψεις και στον προπολογισμό και για σκοπούς εδαφικής ε, συνοχής και υπάρχουν δύο ζητήματα. Με ποιο τρόπο θα προωθούν τόσο μεγάλες διαδρομές. Από δικές μου ενδιαφέρουσες εμπειρίες είδα ότι πρέπει να υπάρχει ένα master plan, ένα γενικό μια γενική σύλληψη για την διαδρομή και μια και βρισκόμαστε στην αρχική φάση προγραμματισμού για τα κονδύλια, θα πρέπει κάποιες περιοχές να έχουν μια κοινή στρατηγική επενδύσεων. Έπειτα πρέπει να εμπλακούν και οι μικρές, οι ελάχιστες, οι κυμεσές επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις στον χώρο της ονομαζόμενης ε, υποδοχής, της ταπεινής υποδοχής, ε, αλλά που είναι τόσο διαδομένη. Μικρές πολιτιστικές επιχειρήσεις, ε, επιχειρήσεις στον χώρο της δημιουργίας που μπορούν να παράσχουν και επιχειρήσεις. Και μετά υπάρχει και άλλο ένα θέμα που έχει να κάνει με, τα, με τις υποχρεώσεις Εκεί μπορούν να είναι πολύ σημαντικές οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και οι δημιουργικές ασχολίες που διατηρούν ζωντανές αυτές τις διαδρομές. Η δάλωση διαδρομή χάνει το νεμά της. Παρ' όλα αυτά θα περιμένουμε τον προπολογισμό 2017 και καλό θα είναι να δώσουμε έμφαση στι εκκλήσει μα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ ένα εκπρόσωπο τη Επιτροπή που θα θέλει και το λόγο, απλώ το ρωτώ. Διότι είτε στον μικρό προπολογισμό που καταφέραμε να προβλέψουμε και που έχει αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Growth, αυτή των διδρομών, 2 εκατομμύρια, νομίζω για 1 εκατομμύριο μόλι, ε, έχουν περικοπεί πάρα πολύ σε σχέση με τι αρχικέ επενδύσει και νομίζω ότι αυτό είναι κρίμα, διότι είναι ένα θέμα που προσελκύει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον. Και έπειτα θα πρέπει να, προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε στη μελλοντική πολιτιστική διπλωματία το θέμα των διαδρομών, διότι μπορούμε να το ε, μεταβάλουμε σε ένα μεγάλο σημαντικό εργαλείο διπλωματική ε, συνομιλία με χώρε που μα ενδιαφέρουν. Αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουμε από κατά νου. Εάν δεν υπάρχουν άλλε παρεμβάσει, θα έλεγα ότι μπορούμε να κλείσουμε εδώ. Σα ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι θα Έχουμε έτσι συναντηθεί και συνομιλήσει. Και ελπίζω οι συνάδελφοι ότι εκτίμησαν αυτές τις τόσο λαμπρές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας δώσατε και όπως είμαστε... Είμαι και μόνιμη συγκέντρια για τη Δημιουργική Ευρώπη. Αυτό είναι ένα θέμα που πραγματικά μου είναι προσφυλέ και θα χαρώ να το παρακολουθήσω. Σα ευχαριστώ λοιπόν και ολοκληρώνουμε την πρωινή μα συνεδρίαση. Θα συνεχίσουμε στι 3 ε, ακριβώ με τη σημαντικότατη ακρόαση για την ένταξη των προσφύγων και των παιδιών τους μέσα της εκπαίδευση και του πολιτισμού. Στις τρεις, Ευχαριστώ πολύ και καλή σας μέρα.